Ladies and gentlemen, let's get started. My name is... ας ξεκινήσουμε. λοιπόν. Πρόκειται για μια ε, ενεργή με, ε, με ανάβραση ε, δραστηριότητα με, με τίτλο Πρόκειται για την Ευρώπη μας. Ας δραστηριοποιηθούμε. Έχουμε δύο ομάδες ε, προσκεκλημένων. Έχουμε 180 λεπτά. Συνήθως έχω μόνο 10 λεπτά κατά τα προγράμματά μου στην τηλεόραση. Έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και είμαστε συνδεδεμένοι με 30 γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 20 γλώσσες χάρη σε όλους τους διερμηνείς που βλέπετε εδώ πίσω και έχουμε επίσης σύνδεση με το Twitter σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και αυτοί που δεν είναι στο γραφείο τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι το hashtag είναι EYC, όπως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών, ή e O, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Φέτος είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά των Πολιτών, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών. Του χρόνου θα έχουμε ευρωεκλογές βεβαίως, όπως ξέρετε. Οπότε έχουμε αυτή την αίσθηση ότι πρέπει να δράσουμε για τους εξή λόγους. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε εκλογές στην Κροατία που θα ενταχθεί πολύ σύντομα στην Ένωση και συμμετείχαν μόνο το 21% των ε, εκλογέων. Στις ε, προηγούμενες ε, ευρωεκλογές είδαμε μια σταθερή μείωση της συμμετοχής των, πολιτών τι θα έχουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να αποδείξουμε σε όλους ε, τους Ευρωπαίους ε, και παρά το ότι έχω αμερικανική ε, προφορά έχω και γαλλικό διαβατήριο και μιλάω πέντε γλώσσες. Πόσοι λοιπόν από τους συμπολίτε μου, τους Ευρωπαίους, θα ψηφίσουν σε ευρωεκλογές, ευρωεκλογές του χρόνου και αν δεν ψηφίσουν τι θα γίνει. Όπως λέγαμε κάποτε ως σύνθημα στον πόλεμο του Βιετνάμ αν γινόταν ένα πόλεμο και δεν πήγαινε κανένα, το πούμε και τώρα. Ε, αν γινόταν εκλογέ και δεν πήγαινε κανένα, δεν ψήφισε κανένα, θα είχαμε πραγματικά υπαρξιακή κρίση. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι μέσω του διαμεσολαβητή, μέσω τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, χάρη σε αυτή τη νέα δυνατότητα που μα δίνει η συνθήκη Λισαβόνα, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την εξουσία και έχουμε ορισμένου ειδήμονε εδώ που θα μα εξηγήσουν πώ μπορούμε να δράσουμε. Ελπίζουμε λοιπόν να αποδείξουμε ότι οι αμφισβητούντες έχουν άδικο. Ναι, μπορούμε να συμμετάσχουμε σε επίπεδο βάσης μέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών, μέσω του διαμεσολαβητή ή κάνοντας αυτό που κάνουμε καλύτερα. Ο καθένας ό,τι του αρέσει. Και αυτό θα σας δείξουμε σήμερα. Να σας παρουσιάσω τους ομιλητές. Αριστερά μου. Ο κύριος Μαρκ Μπερτρό, που είναι διαμεσολαβητής για τη Βαλονία έχει πολλά να μας πει για την ε, Βαλονία, για τα θέματα που αντιμετωπίζει. Δίπλα του είναι η Επίτροπος Vivian Redding, Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνη, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθαγένεια, Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίπλα είναι ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, που είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητή. Εδώ, αριστερά μου, μία έκπληξη, γιατί περιμέναμε τον Μάρτιν Σούλτς πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως ε, εκπροσωπείται από την Ιζαμπέλ Ντουγάν, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ο κύριο Σούλτ προσπαθεί, όπω θα έπρεπε, να έρθει σε επαφή με του πολίτε στην Κύπρο, όπου, όπω ξέρετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δίπλα στην ε, Ιζαμπέλ Ντουγάν είναι η Αλεσάνδρα Μιράμπιλε, που είναι από την ε, αδελφότητα 2020 που αξιοποιεί την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών για να αποκτήσει περισσότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αυτούς τους νέους Ευρωπαίους που θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Έρασμος και άλλα για να σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα από τη χώρα καταγωγής της. Και δίπλα είναι ο Didier Colverts που είναι επικεφαλής ε, της πρωτοβουλίας G1000 είναι μια πρωτοβουλία των ε, πολιτών του Βελγίου που ξεκίνησαν σαν μια τρελή πρωτοβουλία που ήθελαν να πιέσουν ε, να δημιουργηθεί κυβέρνηση στο Βέλγιο όταν δεν είχε δημιουργηθεί πριν από ένα χρόνο. Και ελπίζουμε να ακούσουμε και από αυτού, αλλά και από άλλου που μπόρεσαν να επηρεάσουν τι εξελίξει. Α ξεκινήσουμε με τον κύριο Διαμαντούρο, τον διαμεσολαβητή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Διαμαντούρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρνς, ευχαριστώ σε όλους σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε αυτή τη διαδραστική εκδήλωση με τίτλο «Πρόκειται για την Ευρώπη μας, ας δραστηριοποιηθούμε». Σημειώνω ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013. Έτσι λοιπόν επικεντρωνόμαστε στους πολίτες και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της Ευρώπης και του μέλλοντός της. Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι τους εκπροσώπους πολλών πρωτοβουλειών πολιτών, κινημάτων βάσης και ατόμων που έκαναν καταγγελίες στον Ευρωπαϊκό ε, Διαμεσολαβητή, ε, που όλοι συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο στον να ο στον οποίο ζούμε. Προσβλέπουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούνε ώστε να εμπλακούν στο θέμα της εκδήλωσής μας. Λυπάμαι πάρα πολύ που απροσδόκητα άλλαξε το πρόγραμμα του Προέδρου Σούλτς, πράγμα τον οποίο τον εμποδίζει να παρευρεθεί όπως είχε ε, προγραμματιστεί στην εκδήλωση αυτή. Η παρουσία του στην εκδήλωση αυτή πέρυσι, μαζί με την παρουσία του Προέδρου Μπαρόζο και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Τόρνινγκ Σμιτ, ε, βοήθησε πολύ στην επιτυχία και των προσπαθειών μας να συμμετάσχουν άμεσα οι πολίτες στον ουσιαστικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα για τις συνεχιζόμενες εξελίξεις που επηρεάζουν βαθύτατα τις ζωές και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, με μεγάλη χαρά, πράγματι με μεγάλη χαρά, υποδεχόμαστε την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ιζαμπέλ Ντουραν, η οποία συμφώνησε να βρεθεί σήμερα μαζί μας και ως εκ τούτου εξασφαλίσει την παρουσία του μοναδικού δημοκρατικά εκλεγμένου θεσμικού οργάνου που και που εκπροσωπείται σε αυτή την εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβήτη. Η κυρία Ντουιράν επασύγνωστη για την ενεργό συμμετοχή τη στην ε, κοινωνία των πολιτών και ω εκ τούτου είναι πάρα πολύ κατάλληλη για να λάβει αυτό το έργο. Επίση, είμαστε ευγνώμονε για, την παρουσίαση, για την παρουσία τη και προσβλέπουμε στο να ακούσουμε τι απόψει για τη συμμετοχή των πολιτών στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι, γιατί μα παρήχε την φιλοξενία και στο λαμπρό αυτό κτίριο για την ετήσια εκδήλωση που απευθύνεται σε μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, με την έννοια αυτή θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν βρισκόμαστε μόνο εδώ, αλλά βρισκόμαστε επίσης και σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα γραφεία, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα γραφεία πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε στην Πρατισλάβα, στο Βερολίνο, στην Πράγα και στο Παρίσι, όπως επίσης και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσε. Προσβλέπουμε στο να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσω του Twitter από όλα τα γραφεία πληροφοριών και από όλους όσοι μας παρακολουθούν ε, επιγραμμικά. Ε, είμαι και πάλι πολύ που η, αντιπρόεδρο, η Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ρέντινγκ, βρίσκεται μαζί μας σήμερα και μας τιμά με τη συμμετοχή της σε μια σημαντική εκδήλωση του Γραφείου του Διαμεσολαβητή. Η κυρία Ρέντινγκ είναι στο, στο στην πρώτη γραμμή του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους πολίτες. Στους τελευταίους μήνες έχει ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συναντηθεί με χιλιάδες πολίτες και να ακούσει τα θέματα που τους ανησυχούν. Στη Γερμανία ή στην Ελλάδα βρίσκεται πάντα ε, κάπου για να μιλήσει με τους πολίτες και όχι περί των πολιτών. Ε, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα υποδεχθούμε έναν άλλο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής τον κύριο Μάρου Σεύκοβιτς. Ο κύριος Σεύκοβιτς μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνο για, την, ε, για τις ε, πρωτοβουλίες, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών. Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πολλά για αυτές. Επίσης θέλω να ε, χαιρετήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μάρκ Μπερτρόν, που είναι ο διαμεσολαβητής της Βαλονίας και της Ομοσπονδίας Βαλονίας Βρυξελών, όπως επίσης και τον κύριο Chris Burns από το Euronews, ο οποίος ε, ε, δέχθηκε να συντονίσει τη σημερινή εκδήλωση. Πριν ξεκινήσουμε, να σα πω κάποιε σκέψει μου. Συναντιόμαστε εδώ σήμερα με στο πλαίσιο μιας ε, από τις χειρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, της χειρότερης κρίσης. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μου, όπως και άλλα κράτη-μέλη, σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές ε, διαστάσεις αυτής της κρίσης. Καθημερινά όλο και πιο άσχημα νέα ακούμε, όχι μόνο σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές αγορές, αλλά επίσης για την ε, αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή που έχει σχέση με τα μέτρα λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Ε, όσο σοβαρή κι αν είναι η κρίση για το μέλλον τόσο του ευρώ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει παρατάφτα μια δεύτερη σκοπιά για την κρίση αυτή η οποία πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Πολίτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα όχι μόνο των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα. Ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτό το θέμα κυρίως δεδομένου ότι ένα μέρος αποστολής μου είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη είναι μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και της Ευρωπαϊκής Διοίκησης. Αλλά το ένα είναι να κάθεται κανείς και να περιμένει τις ε, εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνισμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσουν στα προβλήματα αυτά μέσω πρωτοβουλειών και είναι τελείως άλλο θέμα να δράσει κανείς προκαταλαμβάνοντας την κατάσταση αυτή, λαμβάνοντας θετικά μέτρα από μόνος του. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών Πολιτών και των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι πραγματικά σημαντικά ε, βήματα ε, στον μακρύ δρόμο της στήριξης και ενίσχυσης ε, του δικαιώματος των πολιτών να συμμετάσχουν στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνω πάρα πολλές καταγγελίες από πολίτες για προβλήματα στους τομείς αυτούς. Το θεωρώ καλό σημάδι δεδομένου ότι με βοηθούν να ανακαλύψω τα πιθανά μειονεκτήματα της ευρωπαϊκής διοίκησης και να καταλάβω την κατάσταση και να προσπαθήσω ε, να διορθώσω τα προβλήματα. Είμαι πολύ ευτυχής που συνεισφέρω στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών που θα, και ότι αργότερα θα ακούσουμε πώς οι καταγγελίες των διαμεσολαβητή πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Σημερινή εκδήλωση θα μας βοηθήσει να ε, δούμε τι κάνουν οι πολίτες, τουλάχιστον εν μέρη, και να, για να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους και να συνεισφέρουν διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μέλλοντός της. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το επιτύχει κανεί αυτό, Η χρήση των μέσων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω οι, οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών ή η κοινοτοποίηση μεγάλων ομάδων πολιτών για τις ε, πρωτοβουλίες βάσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε αυτή την ε, πρωτοπόρο συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, για να ακούσουμε από τους, τις προτάσεις που θα έρθουν είτε από εδώ από τις Βρυξέλλες ή από τις 30 πρωτεύουσε και πόλει ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν με την ευκαιρία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο όλοι δείχνουμε ε, τα σημαντικά ωφέλη προ του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προέρχονται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τι πολλαπλέ διατάξει τη για την συνεχιζόμενη διαβούλευση και το διάλογο μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Νομική Τάξη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Νικηφόρα να πάμε σε ένα άλλο αλεξικέραυνο. Γιατί και ο νικηφόρος είναι αλεξικέραυνο, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα γίνουν εκλογές του χρόνου. Η Ιζαμπέλ Γιουρό παρακαλώ. Ε, τι θέλετε να πείτε κι εσείς ως αλεξικέραυνο όπως και ο Μάρτιν Σούλτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους. Κύριε Διαμεσολαβήτε, αγαπητέ Νικηφόρε. Κυρίες και κύριοι, και όσοι επίσης από μακριά μας παρακολουθούν ίσως και στη Λευκοσία, στην Αθήνα, στη Μαδρίτη, στη Λισαβόνα. Ίσως ε, δεν έχουν την ίδια διάθεση όπως όσοι είναι εδώ στην αίθουσα. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να μας δείχνει το δρόμο στην πορεία μας, ε, όχι μόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές σε ένα περίπου έτος, αλλά ακόμα περισσότερο για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σωστά ή λάθος ε, σήμερα βλέπουμε ότι χάνουν το ενδιαφέρον τους στην εμπιστοσύνη τους, ε, ίσως όχι τους παλαιότερους αλλά σίγουρα τους νεότερους ε, παρόλο που ο διαμεσολαβητής μας και άλλοι παράγοντες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούν και ξεχωρίζουν όπως θα το πούμε αυτές τις μέρες για να δουν πώς μπορούν να δώσουν ένα κλειδί κατάλληλο Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες η εμπιστοσύνη και είναι τεράστια η δική μας η ευθύνη και κυρίως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε εμά, σε εμάς τους εκλεγμένους, αλλά όσους επίσης εργάζονται για τους εκλεγμένους και όσους εκλέγουν τους εκλεγμένους. Σε ένα έτος ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να είναι εκείνο το παράγον ε, ε, που στην επιλογή των πολιτών θα μπορούσε ίσως να πληρώσει την ύφη εδώ λόγω της κρίσης που σημειώνεται ακριβώς να αντιμετωπιστεί έτσι από πολλούς πολίτες. Βέβαια από τη μια μεριά ο κόσμος εκλέγει, επιλέγει και εκλέγει εκείνος που θέλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και άλλοι που θα απόσχουν, δεν θα ψηφίσουν αλλά επίσης άλλοι που θα ψηφίσουν θυμωμένα, ταραγμένα, ε, με οργή και αυτή η οργή θα μπορούσε να έχει να κάνει με κόμματα που είναι υπέρ ενός νέου εθνικού κεντρικού χαρακτήρα και άλλοι που θέλουν επίσης να φτιάξουν έτσι με τέτοιο τρόπο ε, τα πράγματα που να δείξουν ότι δίθεν σε εθνικό επίπεδο θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζουμε, μέσα στο οποίο ζούμε και στο οποίο θα πρέπει όμως να κινητοποιήσουμε τους πολίτες ε, να καταλάβουν και το κατάλληλο κλειδί που έχουν στα χέρια τους, αλλά επίση και τη σημασία που έχει να δηλώσουν πράγματα, να πούν πράγματα, αλλά και να ακουστούν. Και το να ακουστεί κανείς είναι κάτι που στο ρόλο του διαμεσολοβητή, είτε ενό εκλεγμένου, ακόμα και ενό υπουργού στο Συμβούλιο ή ενό επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το να ακούγεται κανείς είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να απαντήσει και υπάρχουν πάρα πολλέ συναντήσει και διαβουλεύσει με του Ευρωπαίου πολίτε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό είναι να ξέρει κανεί τι θα γίνει με τη γνώμη αυτή. Και πολλέ φορέ κανεί υποφέρει, καταπιέζεται γιατί μια γνωμονή κάτι που πρόσφεραν μια μη κυβερνητική οργάνωση, μια ομάδα πολιτών ή διάφοροι άλλοι φορείς και παράγοντες θα μπει σε ένα κουτάκι, σε ένα σιρτάρι και τελικά δεν ξέρουν σε τι θα εξυπηρετήσει. Για αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών ακριβώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι πολύ νωρίς για να κάνει κανείς μια εκτίμηση και πριν από ένα χρόνο είχαμε στο Στρασβούργο και μια εβδομάδα πριν, αλλά ανοιχτή συζήτηση. Δεν ξέρουμε τώρα από τώρα ακριβώς τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία για γιατί υποφέρει από τι ασθένειε της νεανικές εφηβικές. Έχουμε διάφορα πράγματα που πρέπει να υπογραφούν τον άλλο και η Επιτροπή είναι στην κατάλληλη θέση για να μπορέσει να βελτιώσει αυτό το εργαλείο, αλλά τουλάχιστον θα δούμε εδώ αν με ορισμένε πρωτοβουλίε ευρωπαϊκέ θα μπορέσουμε και με το αίτημα αυτό στην Επιτροπή να επιστρέψει κανεί για ένα ναι ή να όχι για αυτή την πρωτοβουλία, ότι κανεί τη βρίσκει σωστή, καλή και αν όχι δεν είναι ενδιαφέρουσα, σπουδαία, καλή κλπ. Δεν θέλει να την υποστηρίξει, τουλάχιστον να δηλώσει κανείς, να εξηγήσει δημόσια γιατί αυτό. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η συλλογή υπογραφών ακριβώς σχετικά με ένα σχέδιο. Κάτι το δεύτερο, και εδώ θα ήθελα να βοηθήσω φόρο τιμή στο έργο του διαμεσολαβητή. Πολλά και διάφορα έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας σας από την πρώτη εκλογή πριν από 10 χρόνια ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σαν να ήταν χθε. Και το ρόλο που παίξατε στην όλη εξέλιξη αυτή του έργου μέσω της θέσης αυτής και εδώ για τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να υπάρξουν οδημές ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα κείμενα γιατί έγινε αυτό, αυτό δεν συνέβαινε ως παλιότερα και επίσης ε, τα όρια αυτού του νέου δικαιώματος ε, και μας πείσατε ιδιαίτερα για μια κάποια μερεταρρύθμιση, αλλαγή για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση και επίσης μια καλύτερη νομοθεσία, με διάφορες διαβουλεύσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς ακριβώς θα επηρεάζουν τα πράγματα και να δούμε ακριβώς μια νέα ρύθμιση. Και εσείς αυτή την καλή συμπεριφορά την τονώσατε, την ενισχύσατε και πήγατε ένα βήμα παραπάνω με διάφορες αρχές ε, της δημόσιας αυτής υπηρεσίας που θα πρέπει να καθοδηγεί την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που είναι σε επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες και τονίσατε και τη σημασία ότι μια καλή χρηστή διοίκηση δεν είναι απλά και μόνο ένα σεβασμός του δικαίου αλλά πρόκειται για μια αντίληψη γενικά που θα πρέπει να αναπτυχθεί, μια προσέγγιση, ένας τρόπος ζωής απέναντι στους πολίτες Ευρώπης και ότι η διοίκηση είναι στην υπηρεσία των πολιτών και όχι το αντίθετο. Και επίσης εργαστήκατε ιδιαίτερα αποτελεσματικά με διπλωματία, είναι κάτι πολύ σημαντικό, αυτή την καϊκή διοίκηση όπου το συναντήσατε αλλά και διπλωματικά να μην ε, προκαλέσετε μια έλλειψη συνεννόησης ή να σας αγνοήσουν και ε, επίσης επηρεάζει τα πράγματα ακριβώς ανάλογα με την πίθο σας και σίγουρα για τον αντικαταστάτη σας θα αφήσετε σημαντικότατο έργο γιατί σε πάρα πολλές ε, καταγγελίες που απέτησαν την ε, παρέμβασή σας μόνο το 18% δεν ε, είχε μια στο 18% δεν δόθηκε μια συνέχεια και επίσης ένα ειδικό δικαίωμα για μια χρηστή διοίκηση. Βλέπουμε ότι νομικά κάτι τέτοιο είναι δυσμευτικό από το 2009 από την συνθήκη της Σαββόνας και ταυτόχρονα μια νέα νομική βάση το άρθρο 298 της συνθήκης για την οθέτηση νομοθετικών πράξεων για να δούμε ακριβώ να πλαισιώσουμε αυτό το δίκαιο το δικαίωμα και υπάρχουν προσπάθειες εδώ και τρία χρόνια για να δούμε τον τρόπο εφαρμογής αυτού του νέου δικαιώματος η έκθεση Μπέρλεγκερ η οποία συζητείται και καλούμε την Επιτροπή σήμερα να παίξει ακριβώς το ρόλο που της αρμόζει στην όλη αυτή διαδικασία. Και ακόμα κάτι για την πρωτοβολία των πολιτών που είναι ακρογωνίας λήθος για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει με τη συμμετοχή των πολιτών. Και αυτά τα διάφορα παραδείγματα τι μας δείχνουν ότι σήμερα σαφώς η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ακριβώς των εκλεγμένων δεν θα μπορέσει να προχωρήσει χωρίς μια περισσότερη συμμετοχή δημοκρατική είτε μέσω αυτών μεταρρυθμίσεων που μόλις σας είπα αλλά και με νέες μορφές που θα δημιουργηθούν και εδώ βλέπουμε στους συμμετέχοντες διαφορά άτομα και από το Βέλγιο το γη χίλια και ότι υπήρξαν. Ε, ε, διάφορες μορφές συμμετοχής βλέπουμε ότι είναι κάτι αποφασιστική μασία ανάμεσα στου πολίτες. Δεν είναι μόνο μια σχέση με τη διοίκηση και με τους εκλεγμένους και το αντίθετο, αλλά και μεταξύ τους οι πολίτες το συζητούν γιατί έτσι αποφασίζουν και αυτό το πράγμα μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο περίπλοκο είναι ένα πρόβλημα και όταν θέλουμε απέναντι στον λογισμό να δώσουμε τη μάχη μας πρέπει να καταλάβουμε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα και ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί το να προχωρήσει κανείς ε, μαγωγή υγεία είναι πολύ εύκολο. Αυτό στέει, ο άλλο στέει, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το άλλο. Όχι, τα προβλήματα είναι περισσότερο περίπλοκα σε ένα κόσμο όπω το σημερινό και ακριβώς ε, το να λαμβάνεται αποφάσεις, να αποφασίζουν οι πολίτες, ε, ομάδες πολιτών για να μπορέσει κανείς να καταλάβει και να γίνει εμπειρογνώμου κατά κάποιο τρόπο ή τουλάχιστον έμπειρο σε αυτά θέματα όπως και εσείς και εγώ. Έτσι λοιπόν αυτά είναι μέσα και εργαλεία που θα πρέπει να αναπτύξουμε, υπάρχουν ήδη και θα πρέπει σίγουρα να τελειοποιήσουμε και για τον διαμεσολαβητή μάλλον εσείς ο οργανωτής ε, που συμμετέχετε και στο Euronews. Ε, είναι ε, εργάζεστε με πολλές γλώσσες για μια γενική ευρωπαϊκή πληροφόρηση, κάτι βέβαια που είναι πολύ δύσκολο και όσοι μας παρακολουθούν σήμερα σε διάφορες πρωτεύουσε ε, είναι συνηθισμένοι απέναντι σε εθνικά μέσα να αντιδρούν και ξέρουμε ότι τα θέματα δεν θα πρέπει όμως έτσι να αντιμετωπίζονται αλλά να έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα γιατί ακριβώς το εθνικός χαρακτήρας είναι κάπως περιορισμένος, δεν είναι σωστότερος για μια ευρωπαϊκή φύσης απόφαση, για μια νομοθεσία, για μια πρόταση για ένα ψήφισμα. Και πιστεύω ότι αυτή η ανάμεσα πολλά κράτη συνεργασία είναι πολύ δύσκολη και για το Ριορούς και το Άρτε που ξεκίνησε ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία και για οποιοδήποτε άλλη μορφή ε, μεσονημέρωσης ε, από την τηλεόραση, την ε, σημαντικότερη ώρα αναμετάδοσης και για τους αυτούς που θα εκλεγούν. Ελπίζουμε να γίνουν γίνεται καλύτερα και εσείς να οργανώσετε πραγματικές συζητήσεις και στην, ανάμεσα σας πούμε και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επίτροπης κλπ. Μια πλατιά συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να δει ένας Γάλλος ένα Τσέχο ή ένα Φιλανδό. Καλό, θετικό θα είναι. Καλό είναι ένας Γάλλος βέβαια με, είτε με ταυτόχρονη μετάφραση είτε με υπότιτλους να ακούσει έναν άλλο να μιλάει ένα Τσέχο, ή ένα Φιλανδό και να ακουστεί έτσι η Ευρώπη. Ποια είναι η άποψή του κάποιου, κάποιον που δεν είναι από το κόμμα σας όχι μόνο αλλά και από τη δική σας τη χώρα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο αλλά είναι ταυτόχρονα πάντα Ευρωπαίος όπως εσείς. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και έτσι ε, διακόπτει ότι αυτό το αρνητικό παιχνίδι αυτή η Ευρώπη. Δεν μ' αρέσει η Ευρώπη. Όχι, φτάνει πια. Οι ευρωπαϊκέ ακριβώ αποφάσει πώ οικοδομούνται και από του εκλεγμένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μετά από προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επίση και από τι εκλεγμένου των κρατών μελών, από του υπουργού, από του πρωθυπουργού και ηγέτε κρατοκυβερνήσεων και από τα Εθνικά Κοινοβούλιο. Ποιο μιλάει για Ευρώπη στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εσεί απευθύνεστε στου εθνικού βουλευτέ για ευρωπαϊκά θέματα, για να ξέρετε τι κάνει ακριβώ ο υπουργό σα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όμω συναποφασίζετε αποφασίζει. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτόν. Αλλά ο Εθνικό Υπουργό σα προτιμά να μιλάει για περιφερειακά εθνικά θέματα, γιατί έτσι στο εφημεριδούλα την τοπική ε, θα ακουστεί, θα φανεί τι ακριβώ έκανε για κάτι που σα αφορά αμέσω. Αλλά δεν κάνει καμία ενέργεια προ τον Υπουργό του να το ρωτήσει τι ακριβώ κάνετε στην ε, ε, μεταφορέ, στην οικονομία ή οποιοδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε συμβούλιο που αποφασίζουν όμω τρομερά σημαντικά πράγματα νομοθετώντας για 450 εκατομμύρια πολίτες. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν την οπτική γωνία που αντιμετωπίζει το θέμα ο καθένας και η βοήθεια του διαμεσολαβητή και αυτό που γίνεται όπως και φέτος με παρουσία σας και όλοι οι άλλοι που μας βλέπουν από μακριά και μας ακούν θα μπορέσει να κινητοποιήσει ενέργεια των πολιτών και προσπαθώ να σπάσει αυτή την κάπως εύκολη εικόνα μιας κλειστή στον εαυτό της τεχνοκρατικής αλλά ζωνικής Ευρώπης. Εντάξει, εν μέρη αληθεύει, αλλά όχι συχνά, όχι πάντα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αποφεληθούμε αυτές τις δυνατότητες για να ακουστεί μια φωνή έτσι και ελπίζουμε η σημερινή μέρα να αποτελέσει μια ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζουά για την παρουσίασή σας. Βεβαίως, πολλοί Ευρωπαίοι ε, είναι αγανακτισμένοι, έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη τους. Θα θέλαμε λοιπόν σε τοπικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα για να μην υπάρξει λαϊκισμός. Ελπίζουμε του χρόνου να το επιτύχουμε. Η Επίτροπος Vivian Redding, Επίτροπος Δικαιοσύνης Θεμελιδών Δικαιωμάτων, και ηθαγένειας. Νομίζω ότι εσείς ε, φέτος στην Ευρωπαϊκή ε, Χρονιά Πολιτών, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, ακούτε, αφού γκράζεστε τους πολίτες. Τι ακούτε λοιπόν. Καλημέρα σας. Και όσοι είναι παρόντες και όσοι μας ακούνε ηλεκτρονικά. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης που είναι μία από τις πρώτες ψηφιακές συζητήσεις που ε, διεξάγουμε αλλά και για τον τίτλο της εκδήλωσης του. Ε, είναι η δική μας Ευρώπη, ας δραστηριοποιηθούμε. Ενεργοί πολίτες που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, που υψώνουν τη φωνή τους, που παίρνουν πρωτοβουλίες. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους πολιτών. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ε, είναι περίπου 20 ετών τώρα και όταν τους ρωτάμε σε δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις τα δύο τρίτα απαντούν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά το ένα τρίτο μόνο θεωρεί ότι ξέρει τι σημαίνει αυτό. Και νομίζω ότι από αυτό το ένα τρίτο, αν τους ρωτούσαν πιο συγκεκριμένα, μόνο το 10% θα γνώριζε ακριβώς τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και αυτό είναι επειδή στο Maastricht αποφασίσαμε και καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ε, νομισματική ένωση, αλλά η ευρωπαϊκή ηθαγένεια έμεινε μόνο στα χαρτιά. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Σύμφωνα με τις συνθήκες, το δικαίωμα καταγγελίας είναι σημαντικό στοιχείο και γι' αυτό υπάρχει ο διαμεσολαβητής και είναι τόσο σημαντικός. Και δεν είναι μόνο ο διαμεσολαβητής. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. που είναι επίσης μια επιτροπή που ε, δρά, δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και συνεργάζεται με τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Υπάρχει λοιπόν ένα δίκτυο οργανισμών που είναι στη διάθεση των πολιτών. Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο. Τώρα οι πολίτες έχουν επίσης το δικαίωμα να απευθυνθούν γραπτό σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο και έχουν δικαίωμα να λάβουν απάντηση. Λαμβάνω ε, κάθε χρόνο περίπου 5.000 επιστολές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι απαντήσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εργασίας, της ε, γενικής μου διεύθυνσης, των συνεργατών μου. Το πρόβλημα με τις επιστολές αυτές είναι ότι πάνω από τις μισές δεν απευθύνονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Απευθύνονται σε εθνικούς φορείς και δεν λαμβάνουν απαντήσεις σε εθνικό επίπεδο και αυτό τους δημιουργεί απόγνωση. Οπότε η Ευρώπη θεωρείται από πολλούς ε, τελευταία καταφυγή για προβλήματα που δεν ήταν δυνατόν να επιληθούν όπως θα έπρεπε να έχουν επιληθεί, στο επίπεδο που θα έπρεπε να έχουν επιληθεί. Οπότε Ας περάσω στο Ευρωπαϊκό Έτος ε, Πολιτών. Γιατί αποφασίσαμε να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία. Να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί το αποφασίσαμε. Γιατί διαπιστώσαμε ότι μόνο το 1 τρίτο των πολιτών μας θεωρεί ότι παίζει ρόλο η φωνή τους. Οπότε αυτό με φέρνει κατευθείαν στην ερώτηση που έθεσε και η κυρία Ντουρό. Διότι οι πολίτες δεν έχουν το αίσθημα ότι μετράει ο λόγος τους ότι έχει αποτέλεσμα. Εάν δεν θεωρούν ότι έχει αποτέλεσμα ο λόγος τους, δεν θα πούν τίποτα. Δεν θα πούν τίποτα στην καθημερινή τους ζωή και ίσως ε, να μην προσέλθουν και στις κάλπες. Ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το 21% στις ευρωεκλογές ε, της Κροατίας. Και για να καλύψουμε αυτό το κενό, για να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι ναι, μετράει η φωνή σας, δεν χρειάζεται να κάνουμε μακροσκελής ομιλίες, διότι έχουν μπουχτίσει από τέτοιες ομιλίες οι πολίτες. Μπορεί να γίνει αυτό μόνο. Αυτό που οι πολιτικοί δεν ξέρουν να κάνουν. Να το βουλώσουν και να ακούσουν τι τους λένε οι πολίτες και να ανταποκριθούν. Και γι' αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε τους διαλόγους με τους πολίτες. Έχουμε διοργανώσει πολλούς, σε πολλά μέρη. Και, συνειδητότατα, προσπάθησα να οργανώσω αυτούς τους διαλόγους εκεί που υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο πρώτος τέτοιος διάλογος έγινε στην Νότια Ισπανία, τα Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία κλπ. Είχαμε εκατοντάδες πολίτες ε, που για ώρες απλώς έκαναν ερωτήσεις και λάμβαναν απαντήσεις. Δεν γινόταν καμία ομιλία. Και τι μας ε, καταδεικνύει αυτό. Πρώτα απ' όλα εκπλήσονται οι πολίτες. Λένε πρώτη φορά έρχεται να μας ακούσει ένας πολιτικός. Δεν μας έχει συνηθίσει η πολιτική σε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, περίμενα βέβαια να ακούσω ότι η Ευρώπη δεν τα πάει καλά, η Ευρώπη δεν ε, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Όχι. Το αντίθετο διαπίστωσα. Θέλουν περισσότερη Ευρώπη. Και δεν τους ενδιαφέρει για το ποιος οργανισμός ποιο θεσμικό όργανο θα λύσει το πρόβλημα. Θέλουν απλώ να επιληθεί από κάποιον. Όλη αυτή λοιπόν η θεσμική συζήτηση που θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική για μα δεν είναι για του πολίτε. Θυμάμαι στο Βερολίνο. Είχα ε, ε προετοιμαστεί να μιλήσω για τα αγκουράκια, για άλλα θέματα γλόμπων, για μικρά θέματα και να πω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εμπλακεί σε τέτοια θέματα. Να σα δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα αυτό που άκουσα. Μία κυρία είπε έχω προβλήματα στο σχολείο με το παιδί μου. Ε, μου είπε λοιπόν, κυρία Επίτροπε, εσεί δεν πρέπει να λύνετε τα προβλήματα. Λύστε το. Ε. Προσπαθούσα να εξηγήσω στην ε, κυρία αυτή ότι με βάση τι ευρωπαϊκέ συνθήκε τα προγράμματα σπουδών ε, των σχολών είναι θέμα που λόγω της επικουρικότητας πρέπει να το εντοπίσουν τα κράτη. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αλλάξουμε την συνθήκη. Και ξέρετε τι μου απάντησε. Ελίστε το πρόβλημα αλλάζοντα τι συνθήκε. Εξήγαγα θαυμάσια διδάγματα. Ο περίπλοκος τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να λαμβάνουν απλή απάντηση στις απλές ερωτήσεις τους και κάποια δράση. Κάντε κάτι μας λένε. Κάντε κάτι. Γι' αυτό ξεκινήσαμε την προετοιμασία των διαλόγων με τους πολίτες πέρυσι το Μάιο. Μέσω της πρώτης προσπάθειας ε, να λάβουμε αντίδραση των πολιτών μέσω του διαδικτύου. Λάβαμε 12.000 ε, παρατηρήσεις όλες οι ε, παρεμβάσεις ήθελαν περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενοποίηση και περισσότερη άμεση δράση, χωρίς γραφειοκρατία. Η έκθεση λοιπόν που παρουσίασε για τις επιθυμίες των πολιτών ήταν ένας κατάλογος συγκεκριμένων θεμάτων όπου έπρεπε να δράσουμε. Συστάσεις δράσης και από τις 25 συστάσεις αυτές που προτείναμε πριν από δύο χρόνια, 24 έχουν εφαρμοστεί. Θα υπάρξει επίσης μια νέα τέτοια έκθεση ε, τον επόμενο μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που μας είπαν οι πολίτες, όχι μόνο μέσω των διαλόγων που διοργανώσαμε, αλλά και μέσω των 5.000 επιστολών που λαμβάνουμε ετησίως και μέσω του ενός εκατομμυρίου ερωτήσεων που θέτουν μέσω του Europe Direct Ξέρουμε τι ενδιαφέρει τους πολίτες. Δεν θέλουν γραφειοκρατία. Θέλουν να διευκολυνθούν στην ελεύθερη διακίνησή τους. Αυτά είναι από τα σημαντικότερα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Φέτος λοιπόν θα διατυπώσω 12 συγκεκριμένες προτάσεις που θα εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να πούμε στους πολίτες ναι, μετράει ο λόγος σας, ναι, ακούμε τη φωνή σας, διότι λαμβάνουμε τις προτάσεις σας οι οποίες καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι λόγια, όχι μπλα μπλα, μια συγκεκριμένη προσπάθεια, ε, πρόβλημα, επίλυσή του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι πολιτικοί να καταδείξουν ότι ακούνε τους πολίτες και ότι εξηγούν τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και τους εξηγούν επίσης σε ποιο επίπεδο μπορεί να εξευρεθεί λύση για κάποιο θέμα. Γιατί ορισμένε φορέ ε, κάποια προβλήματα μπορούν να επιληθούν σε τοπικό ή περιφερειακό. Δεν είναι ανάγκη να επιλύονται όλα τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Έτο των Πολιτών δεν είναι απλώς ε, πείραμα εργαστηριού, αλλά πολιτική αναγκαιότητα, ιστορική ευθύνη. Όλοι οι επίτροποι συνεργάζονται με τους ευρωβουλευτές, συνεργάζονται με τους υπουργούς ε, με τους δημάρχους για να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Και νομίζω ότι έχουμε τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Ελπίζω αυτό να επηρεάσει και την προεκλογική εκστρατεία, ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη αλληλεπίδραση σε όλα τα επίπεδα και ελπίζω να επηρεάσει και κάτι άλλο, την προετοιμασία των επομένων συνθήκων, ούτως ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε. Αλλά όχι ε, πάλι με τον ε, συνήθι στο παρελθόν τρόπο. Δηλαδή εκλέγαμε κάποιους σοφούς οι οποίοι συζητούσαν για να καταλήξουν σε λύσεις και οι λύσεις αυτές αναγγέλλονταν στους πολίτες λέγοντάς τους ε, έτσι θα γίνουν τα πράγματα είτε σας αρέσει είτε όχι. Τώρα πρέπει να συμμετάσχουν εξυπαρχείς οι πολίτες στη συζήτηση τροποποίηση των συνθήκων. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε τι περίπου θα μα απασχολήσει μέχρι να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε διατυπώσει. Ούτω ώστε οι πολίτε να συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία τροποποίηση των συνθήκων. Και όταν θα πρέπει να ψηφίσουν, για παράδειγμα, σε ένα δημοψήφισμα, να γνωρίζουν ήδη περί τίνος θα ψηφίσουν. Γιατί είχε συμπεριληφθεί η άποψή του στη διατύπωση των θεμάτων επί των οποίων θα ψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Ρέντινγκ, ε, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Και σημειώνω ότι ήσασταν ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, άρα έχετε συμμετάσχει πολύ ενεργά 89 ε, και 92 σε μια περίοδο κλειδί, όπου ελέγχαμε πως θα εφαρμοστεί η συνθήκη του Μαστρίτ που παραλίγο δεν περάσει. Ας περάσουμε τώρα σε κάποιον ο οποίος έχει μεγάλη σχέση με τις πρωτοβουλίες των πολιτών, μία προσπάθεια που προσπαθεί να ε, ε δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση των ε, νέων μας. Η Αλεσάνδρα Μιράμπιλε λοιπόν θα σας εξηγήσει πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ομάδα πρωτοβουλίας της. Όπως είπα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες Υπάρχουν ακόμη ε, δυσχέρειες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί στον τρόπο λειτουργίας. Είναι λοιπόν ένα πείραμα αυτό με την ε, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών. Πρέπει να αναφέρουμε αυτά τα αρχικά και δεν μας αρέσει να αναφέρουμε αρχικά. Τώρα λοιπόν ε, οι ομιλητέ μας. Η Γκούντι Γκάτεσμεν σημειώνει εδώ προσπαθώ να δω ε, από τον τρόπο με τον οποίο ε, μοιάζει να αντιδρά εάν έχουμε tweet ενδιαφέροντα ήδη από αυτούς που μας ακούν και από το κοινό βεβαίως και από όσους μας ακούν ε, μέσω του web streaming στον ιστότοπο του διαμεσολαβητή αν έχετε ερωτήσεις, αν έχετε σχόλια Α, βλέπω ότι, βλέπω ότι το tweet λαμβάνει, λαμβάνει συνεχώς καινούργια tweet. Σας είπα το hashtag είναι EYC 2013 EO στα αγγλικά όλα αυτά. Παρακαλώ στείλτε μας όσα περισσότερα tweet γίνεται. Λοιπόν, η Αλεσάνδρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωπαίδε Διαμεσολαβητή, κύριε Διαμαντούρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή μου που απευθύνομαι σε αυτό το διακεκριμένο κροατήριο σήμερα. Θα είμαι πολύ σύντομη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διάδρασης και υποβολής όσο το δυνατόν περισσότερων ερωτήσεων. Θα σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η Αδερφότητα 2020 και γενικώ τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της λύσης της ε, Τρέχουσα οικονομική κρίση, δεδομένου ο τίτλος μας είναι να βοηθήσουμε στην επίλυση τη οικονομική τρίτης, ε, κρίσης. Είναι κάτι που σχεδόν μας φοβίζει ω ερώτημα και πραγματικά η δική μου θα είναι μια πολύ περιορισμένη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση που αφορά την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση και όλα τα σχετικά με αυτήν θέματα. Συγκεκριμένα, αυτό το οποίο παλεύουμε στην για το οποίο παλεύουμε στην εκστρατεία μας είναι να συγκεντρωθούν περισσότεροι πόροι, το 3% του ευρωπαϊκού προπολογισμού ε, που θα πρέπει να πηγαίνει στα προγράμματα ανταλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα από τους, ε, τους σκληρούς αγώνες στο θεσμικό επίπεδο, πιστεύουμε, εμείς η Επιτροπή Πολιτών της Αδερφότητας 2020, πιστεύουμε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να έχουν την εμπειρία του τι ακριβώς σημαίνει η Ευρώπη για αυτούς και να υποφεληθούν από τα, από τα προγράμματα κινητικότητας που προσφέρει η Ευρώπη. Επίσης, γενικότερα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψει τις προσπάθειές της για την ολοκλήρωση στο επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών. Επειδή λοιπόν το 2013 είναι το έτος Ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγμα που σημαίνει ενεργό συμμετοχή, ενεργό δέσμευση των πολιτών. Επιπλέον η αυξημένη κινητικότητα θα έχει και θετικά αποτελέσματα από οικονομική άποψη επίσης, δεδομένου ότι θα ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και θα μειωθεί η ανεργία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κυρίως η ανεργία των νέων που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα όπως όλοι γνωρίζουμε. Ε, σχετικά λοιπόν θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε η, κυρία, ε, η, καθηγήτρια Σοφία Κοράντη, η γνωστή Μάμα Εράσμους, σχετικά με αυτό το έτος 2013 και που έχει σχέση και με αυτό που κάνει η κυρία Ιζαμπέλ Ντουράν και την ευχαριστώ για τη συμμετοχή της. Όταν λοιπόν μιλούσε για τα ωφέλη που, έχουν, που έχει η συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παθιασμένο αλλά και πολύ πιστικό τρόπο είπε ότι τα προγράμματα αυτά γενικότερα αλλά και το πρόγραμμα Εράσμους πιο συγκεκριμένα δεν ε, αποτελεί μόνο ένα τρόπο να ε, έχει κανείς την εμπειρία για την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης, αλλά και είναι ένας τρόπος προς την αγορά εργασία. Και ως εκ τούτου αυτό προσφέρει μια σημαντική προστιθέμενη αξία στα βιογραφικά σημειώματα των νέων καθώς αυτοί προσπαθούν να βρουν μια κανονική δουλειά και όχι ε, απλήρωτες ή κακά πληρωμένες και αμοιβόμενες μαθητείες. Όλοι γνωρίζουμε το φαινόμενο αυτό πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, με βάση την προσωπική μου εμπειρία, επειδή έζησα στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, πρέπει να προσθέσω ότι το να ζει κανείς στο εξωτερικό αποτελεί μια εμπειρία που σε μαθαίνει πολλά, σου αποκαλύπτει πολλά, σε βοηθά να διαμορφώσεις την προσωπικότητά σου, να, να έχεις μια άλλη αντίληψη της ζωής και να σκέφτεσαι ως ελεύθερο άτομο. Κάτι που δεν είναι τόσο απολύτως δεδομένο στη, ακόμα και στις ελεύθερες, δημοκρατικές, φιλελεύθερες κοινωνίες μας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι όταν συζητάμε για το πρόγραμμα Εράσμους και τα προγράμματα ανταλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η προσέγγιση μας να είναι πιο ολιστική. Να μην τα αντιμετωπίζουμε μόνο ως διακοπές που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία, την Κύπρο, τη Μάλτα ή και στο Βέλγιο για αυτούς που θέλουν πολύ να, να βρίσκονται εδώ. Και για να μιλήσω πιο σοβαρά, πρέπει να υπογραμμίσω ότι παρότι δεν θεωρούμε ότι ο ένας, ο, ότι εμείς οι, οι άλλοι συνομιλητές μας είναι απλώς ε, αγαθοί στα θέματα της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει η Ευρώπη ένα καλύτερο μέρος για όλους μας. Βρισκόμαστε σε περίοδο βαθύτατης κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική και χρηματοπιστωτική. Είναι κρίση δημοκρατίας, κρίση εμπιστοσύνης στη διακυβέρνηση και στα θεσμικά όργανα όπως είπε η κυρία Ζαμπέλ Ντουράν και, ε, και το οποίο επεσήμανε και ο κύριος Διαμαντούρος. Στην περίοδο αυτή της κρίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες. Στην περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικό οι επενδύσεις στους νέους Ευρωπαίους, το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει η Ευρώπη, να είναι προτεραιότητα. Όχι μόνο λοιπόν να γίνονται επενδύσεις στη γεωργία, στα διαρθρωτικά ταμεία και στα ταμεία συνοχής, και αυτά είναι πολύ σημαντικά βεβαίως, αλλά και επενδύσεις σε δραστηριότητες ε, του μέλλοντος, όπως ε, φυσικά η παιδεία. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές προκλήσεις ε, που έχουμε τώρα, αν θέλουμε να ε, προσχωρήσουμε στην ε, οικονομική ανάπτυξη που είναι κάτι που απασχολεί την Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα αποτύχουμε και εξίσου θα αποτύχουν αργότερα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι λοιπόν μπορεί μια μεγάλη επιτυχία να δημιουργηθεί όχι μόνο με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης και της Δημοσιονομικής Ένωσης αλλά και με το να μπει το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας στην πράξη και να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των προγραμμάτων ανταλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει αυτό πράξη. Οι, οι νέοι Ευρωπαίοι, οι νέοι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνει για αυτούς η Ευρώπη. Βεβαίως, για να επιτευχθούν αυτά, πρέπει να δεσμευτούμε, να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο να δουλέψουμε για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα είναι πιο δεκτικό στην συμμετοχική δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών ελπίζουμε σε αυτό το τομέα θα πετύχουν. Έτσι λοιπόν σας ενθαρρύνω βεβαίως να ενισχύσετε την συμμετοχική δημοκρατία και βεβαίως να πάτε στο διαδίκτυο για να υπογράψετε τη δική μας πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Περιμένω ε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, Αλεσάνδρα. Αντιλαμβάνομαι πώς ε, σε απασχολεί αυτό το θέμα που πολλοί αποκαλούν δημοκρατικό έλλειμμα και πώς σήμερα θα το περάσουμε μέσω των αναφορών, μέσω των ε, ε, πρωτοβουλειών της βάσης. Έχουμε και έναν άλλο διαμεσολαβητή σήμερα, τον Μάρκ Μπερτράν, ο οποίος είναι διαμεσολαβητής της Βαλονίας. Θα έχεις πάρα πολλές ιστορίες να μας πεις, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε ε, διαμεσολαβητή, ε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρο του Βουλίου, αγαπητοί φίλοι που είστε εδώ παρόντες και μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που ε, έχουμε στη διάθεσή μας και εκτός του κτίριου. Καταρχάς, να ξαναθέσω το πλαίσιο του αιτήματο που μετέθηκε να πάρω το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Να υπενθυμίσω το πλαίσιο ότι θέλουμε να αφαιρωθούμε στους πολίτες και να συμβάλλουμε στον τρόπο που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, μου ζητήθηκε να παρέμβω για το θέμα συμβολή στην επίλυση της οικονομικής κρίσης. Και πιο συγκεκριμένα να σας μιλήσω για την εμπειρία μου ως ε, κοινοβουλευτικός και θεσμικός διαμεσολαβητής εδώ στο Βέλγιο δεν φιλοδοξώ ως διαμεσολαβητής να απαντήσω διαρθρωτικά στον τρόπο και στις λεπτομέρειες επίλυσης της οικονομικής κρίσης. Προφανώς, παρόλα αυτά, μέσω της δράσης του διαμεσολαβητή που θα σας παρουσιάσω σύντομα μπορούμε πιστεύω να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε αυτούς που θίγονται απευθείας από την κρίση. Η διατήρηση και η πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πραγματικό συσύφιο έργο που ξαναρχίζει συνέχεια και ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Εάν έχουμε καμιά φορά την ψευδέστηση ότι έχουν σημειωθεί μεγάλες πρόοδοι, ο χρόνος, αυτός ο καταστροφέα μύθων επενθυμίζει πολύ σύντομα την πραγματικότητα και πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτή η διαπίστωση διατυπώθηκε το 1996 στο Στρασβούργο από την πρόεδρο της Διακυβερνητική Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. δυστυχώ ισχύει ακόμη σήμερα το διάταγμα που δημιούργησε την υπηρεσία ε, του διαμεσολαβητή τη Βαλονία και τη Ομοσπονδία Βαλονία Βρυξέλλε δεν έδωσε εκπεφρασμένα ω πρώτο καθήκον του διαμεσολαβητή τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελινών ελευθεριών των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, μέσω τη δράση του, ο διαμεσολαβητή συμβάλλει πολύ συγκεκριμένα. Ο ρόλο μα είναι να ελέγχουμε την δράση τη διοίκηση, τη σχέση τη με του πολίτε να ελέγχουμε την κάκο διοίκηση και τις δυσλειτουργίες της διοίκησης. Να ε, μπορεί να ε, συμφιλιώνονται οι πολίτες με τη διοίκηση και έτσι να επανέρχεται ή να ενισχύεται η εμπιστοσύνη τους στην ε, διοίκηση και στην κυβέρνησή τους. Αυτό σημαίνει ότι η δράση μου έχει στόχο τις καθημερινές δυσχέρειες των πολιτών έναντι των δημοσίων υπηρεσιών, που θεωρούνται από τους πολίτες οι απαιτήσει τους ιδιαίτερα βαριές, ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τόσα προβλήματα. Όπως το περιέγραφε ε, πρόσφατα ο Γάλλος ε, ε, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλες οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα αιτήματα ικανοποιούνται. Μερικοί θεωρούν ότι είναι θύματα δυσλειτουργίας ή σφάλματος, αλλά αυτό δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, στόχο μα και αποστολή μα είναι να είμαστε μία οδό πρόσβαση δικαιωμάτων για αυτού που δεν καταφέρουν να γίνει ακουστή η φωνή του και να δώσουμε πάλι ανθρώπινο χαρακτήρα στη σχέση μεταξύ του πολίτη και των δημοσίων αρχών. Αντιμετωπίζοντα παράλληλα τι διαμαρτυρίε εκείνων που απευθύνονται σε εμά και κάνοντα προτάσει, ε, τροποποίηση στο Κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση, έχοντα ε, διαπιστώσει εμεί οι ίδιοι τι δυσλειτουργίε ή τα επεισόδια διακρίσεων. Έτσι, ε, υπερασπίζοντας τον πολίτη κατά της ε, κακής λειτουργίας της διοίκησης, ο διαμεσολαβητής συμβάλλει, όπως όλοι οι διαμεσολαβητές, ευρωπαϊκή, ε, εθνική, περιφερειακή συμβάλλει στην προστασία και πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, όταν παραγνωρίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και ακριβώ αυτή η τελευταία διάσταση υπάρχει και στον τίτλο και στη λειτουργία του διαμεσολαβητή σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε αποκαλείται υπερασπιστή των δικαιωμάτων στη Γαλλία, προστάτη των πολιτών στο Κεμπέκ, υπερασπιστή του λαού στην Ισπανία. Και αυτά που θα σα αναφέρω τώρα θα το αποδείξουν. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το άρθρο, ένα άρθρο του συντάγματό μα, λέει ότι ο καθένα έχει δικαίωμα να διεξάγει μια ζωή που να είναι σύμφωνα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και ο νόμος πρέπει να ε, εγγυάται, λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, ανάλογε υποχρεώσει, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και να καθορίζει τι συνθήκε άσκησή των. Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην εργασία και στην ελεύθερη επιλογή επαγγελματική δραστηριότητα, ούτω ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη και πιο ασφαλή εργασία. Επίση, να υπάρχουν δυνατότητε καλών συνδικών εργασία, να υπάρχει δυνατότητα διαβούλευση και συλλογικών διαπραγματεύσεων, δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, στην προστασία τη ε, ε, υγείας και στην κοινωνική, ιατρική και νομική βοήθεια. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή στέγαση, το δικαίωμα ενός ε, υγιούς περιβάλλοντος, το δικαίωμα άσκησης των πολιτιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η αποτελεσματικότητα αυτών των δικαίων σημαίνει παρέμβαση και συμπληρωματική δράση της νομοθετικής εξουσίας. Έτσι, στη χώρα μου, στα διάφορα επίπεδα εξουσίας, έχουμε την υποχρέωση να ασκούμε ουσιοδός αυτές τις προδιαγραφές που τα περισσότερα είναι δικαιώματα των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά, οι κοινοφελείς οργανισμοί και οι διοικήσει στις σχέσεις τους με τους πολίτες δεν, εάν λοιπόν δεν εκπληρώνουν ή εκπληρώνουν λάθος ε, το καθήκον τους, χρειάζεται και αιτιολογείται πλήρως η παρέμβαση του διαμεσολαβητή. Αποτέλεσμα είναι ότι βοηθώντας τους πολίτες που τα δικαιώματά τους όσο αφορά τη στέγαση, την υγεία, το περιβάλλον και την πολιτιστική δραστηριότητα δεν θα υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν γίνει σεβαστά, βοηθώντας τους να βρουν το δίκαιο τους, ο διαμεσολαβητής συμβάλλει στην προστασία και τον σεβασμό των θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Euh? Please bear with us. Please bear with us. Παρακαλώ περιμένετε λίγο. Ελπίζουμε ότι είναι απλώς άσκηση ή λάθος και αυτοί που είναι, μας ακούνε εκτός κτηρίου, ε, πάρετε συναγερμός και ελπίζουμε να επιλυθεί το πρόβλημα. Παρακαλώ, περιμένετε. Α, σταμάτησε, ωραία. No, we didn't stage this. όχι, όχι, δεν, δεν είναι κάτι που το είχαμε σκηνοθετήσει. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπέτραν. Λοιπόν, θα τελειώσω λέγοντας ότι έτσι ο διαμεσολαβητής ε, συμβάλλει στην, ε, στο, στην, στο συμβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων και ο διαμεσολαβητής ούτως ή άλλως ε, λαμβάνει πολλά παράπονα από πολλούς συγκεκριμένους πολίτες που είναι οι πιο ευάλωτοι. Είναι αυτοί που στην κοινωνία μας αποκαλούμε... Please stand by. Ah, All right. Λοιπόν, συνεχίζω. Στην κοινωνία μας λοιπόν πρέπει κυρίως να προσέξουμε μια κατηγορία πολιτών, αυτούς που αποκαλούμε οι Αυτοί που έχουν αποκλειστεί από την εργασία, από τη στέγαση ή από την περίθαλψη. Αυτοί που δεν μπορούν πια να πληρώσουν τους λογαριασμούς ε, νερού, φυσικού αερίου ή ακόμη και ηλεκτρισμού αυτοί που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, τα δίδακτρα για τα παιδιά του. Το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγαση, το δικαίωμα προστασία υγεία είναι θεμελιώδη δικαιώματα. You stand by once again. Okay. Okay. For, for one minute or two maximum. Je Λοιπόν, αναφέρω και πάλι τον κύριο Μποντή. Η σημερινή κρίση ε, ε, αυξάνει τι εντάσει και στι σχέσει μεταξύ των πολιτών, οξύνει τι διαμάχε και οθεί εκείνου που είναι σε ήδη σε ανασφαλεί συνθήκε σε ε, δράσει αγανάκτησης και απόγνωσης. Αλλά δεν, μόνο, δεν φταίει μόνο η έλλειψη πόρων. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Πολλοί πολίτε μας είναι ευάλωτοι λόγω της σκληρότητας της κοινωνίας, της σκληρότητας των συστημάτων. Η τυφλή εφαρμογή κανονισμών, η έλλειψη διαλόγου, η έλλειψη διαφάνειας, η περιπλοκότητα των διοικήσεων ή των οργανισμών μας οδηγούν πολλές φορές σε ένα συνέστημα δίκαια άδικα ότι αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας αδιαφορία και αδικία. Επειδή απευθύνονται σε αυτόν οι περιθεροποιημένοι, ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να βοηθήσει καθημερινά τους συμπολίτε του να διαμορφώσει μια πιο ανθρώπινη και άμεση σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες και μέσω αυτού του τρόπου να συμμετάσχει στην πάλη κατά όλων των μορφών διακρίσεων. Η παρέμβασή του ε, είναι αναγκαία στις σημερινές συνθήκες αυξανόμενης φτώχειας του πληθυσμού και διακοπή παροχή υπηρεσιών, νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, ε, κακή ε, συντήρηση των κοινωνικών κατοικιών κτλ. Ο διαμεσολαβητή ακούει τα άτομα. Είναι μια σημαντική αυτή φάση, όπω ήδη υπόθηκε. Ο διαμεσολαβητή είναι ο εκπρόσωπο των πολιτών έναντι των. Προσπαθεί να ε, βοηθήσει από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να προτείνει στη δίκηση μέτρα και μεταρρυθμίσεις της ε, συμφιλίωσης, αποκατάστασης αδίκων καταστάσεων και κατάδειξης ε, δυσλειτουργιών, ο διαμεσολαβητής είναι παράγων κοινωνικής ειρήνης και συμβάλλει στην διατήρηση με αποτελεσματικό τρόπο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο αείμνηστος Ζακ Πελτιέ, που ήταν ε, διαμεσολαβητής της Γαλλικής Δημοκρατίας, είχε πει «Η διαμεσολάβηση αντιμετωπίζει τον αποκλεισμό στην καθημερινή λειτουργία των διαμεσολαβητών. Ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου τη Ομοσπονδία Βαλονία Βρυξέλλες πρόσφατα απευθύνθηκε στου περιφερειακού διαμεσολαβητέ Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας αυτό το όραμα και προοπτική του ρόλου. Αντιμετωπίζουμε μια οικονομική και κοινωνική κρίση χωρί προηγούμενο. Στην Ευρώπη εξαπλώνονται οι αμφιβολίες, εξαπλώνονται στον πληθυσμό. Σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία ο διαμεσολαβητή μπορεί να είναι προπύργιο τη δημοκρατία, να βοηθήσει τι κυβερνήσει, να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών χάρη στο ρόλο διαμεσολάβησης διαφορετικών απόψεων, προστασίας των πολιτών και ενίσχυσης της σωστής διοίκησης. Όμως ε, δεν πρέπει οι πολίτες να εφησυχάζουν. Αντίθετα, πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη βελτίωση της καλής διακυβέρνησης μέσω της συμβολής μας. Αυτό σημαίνει να δεσμευθεί να ασκεί ο ίδιος έλεγχος στη διοίκηση, ούτω ώστε η ατομική του διαμαρτυρία να βελτιώσει τον κανόνα. Αυτή η αντίληψη του ρόλου τους υποστηρίζεται και εφαρμόζεται από πολλούς διαμεσολαβητές κυρίες και κύριοι. Προσπάθησα να σα αποδείξω ότι ο διαμεσολαβητή μέσω τη καθημερινή του δράση κάνει ό,τι μπορεί, ούτω ώστε η χιονοστιβάδα παθροπιά να μην τα καταστρέψει ε, όλα και να μην καταστρέψει ό,τι έχουμε ήδη επιτύχει και προτείνει. Ο σύσφο, ελευθερωμένο από την καταδίκη των Θεών, θα μπορέσει μια μέρα να φτάσει στην κορυφή του όρου, ε, ε, ε, αναρωτιόταν η κυρία Λεϊτάου μέσω των, οργανώσεων, των ε, εκδηλώσεων που οργανώνεται τώρα, κύριε ε, Διαμαντούρε, ελπίζουμε να υπάρξει ε, συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες κρίσης να ανεχόμεθα τον αποκλεισμό, την ανεργία. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπερτράν. Λοιπόν, μας λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα στο σύστημα, το οποίο φτάνει μέχρι τα μηχανήματα, προσπαθούν ε, να το αντιμετωπίσουν. Ε, λοιπόν, σας παρακαλώ κάντε υπομονή, ελπίζουμε να ήταν η τελευταία φορά που χτύπησε ο συναγερμό. Εν πάση περιπτώσει, μας τελειώνει πολύ γρήγορα ο χρόνος του πρώτου αυτού ε, τραπεζιού. Οπότε περνάμε γρήγορα στον Didier Καλουβέρτ που εκπροσωπεί την ε, κίνηση Βέλγων πολιτών G1000. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την οργάνωση της εκπληκτικής αυτής εκδήλωσης. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους παριστάμενους για που θα παρακολουθήσουν αυτή τη σύντομη παρουσίαση ε, για την πρωτοβουλία G1000 Υπάρχει και κάποια παρεμβολή όπως ακούτε. Η, το G1000 ήταν μια πρωτοβουλία πολιτών που έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ στις Βρυξέλλες όπως και πολλές άλλες πρωτοβουλίες ε, και εκδηλώσεις για, τα, για τις οποίες ακούσαμε πολλά σήμερα. Το G1000 δείχνει την εξαιρετική δέσμευση των απλών πολιτών στην, για τη δημοκρατία τους. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν εντυπωσιακό. Συγκεντρώσαμε 704 τυχαία επιλεγέντες, απλούς Βέλγους πολίτες και από τις δύο γλωσσικές ομάδες, τις τρεις γλωσσικές ομάδες και τους ζητήσαμε να συζητήσουν σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Αυτοί ήταν πολίτες που πολύ συχνά θεωρούνται ότι είναι πολιτικά αδιάφοροι και ε, απαθείς και ότι δεν εμπιστεύονται την πολιτική. Αλλά ταυτόχρονα αυτό έδειξε ότι οι πολίτες με προθυμία δέχτηκαν να μείνουν επί μια μισή μέρα που ήταν αργία για να συζητήσουν αυτά τα ε, ζητήματα που αφορούσαν όλους. Το G1000 πέτυχε κάτι το οποίο στο Βέλγιο θεωρεί το αδύνατον και ορίστε κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία. Βάλαμε ένα πολύ μακροσκελές μανιφέστο στο διαδίκτυο και μέσα σε 10 μέρες το υπέγραψαν 10.000 πολίτες. Το διάβασαν και το υπέγραψαν. Σε τρεις μήνες ε, από μια ομάδα 7 θελοντών ε, που συνεδρίαζαν γύρω από ένα τραπέζι κουζίνας. Φτάσαμε στο... Α, με συγχωρείς Διτιέ, λέει ο συντονιστής, πρέπει να εκενωθεί το κτίριο. Αυτοί οι οποίοι μας ακούν ε, διαδικτυακά να ξέρουν θα επιστρέψουμε. Πρέπει να εκενωθεί το, το κτίριο. Ευχαριστώ πολύ.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 And Λοιπόν, επανερχόμεθα. Επί 500 ημέρε δεν είχαμε κυβέρνηση στο Βέλγιο και δεν μπόρεσαν να βάλουν τα προβλήματά του στην άκρη. Τελικά, μια μέρα του Νοεμβρίου διαπιστώθηκε ότι ακόμα και οι βαθύτατες συγκρούσει και διαφορέ μπορούν να ξεπεραστούν. Έδειξε την αντοχή τη δημοκρατία, έδειξε ότι οι πολίτε μπορούν να δουν κάτι παραπέρα από τη δική τους άποψη και να προτείνουν λύσεις ακόμα και όταν οι συγκρούσεις είναι βαθύτατες. Θα ήταν καλό ίσως στο σημείο αυτό να επισημάνω κάποια από τα παραδείγματα της ριζοσπαστικής σκέψης των πολιτών πρότειναν καταρχήν τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως ο Tobin Tax, πρότειναν τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας με τη δημιουργία ενός ενιαίου βασικού εισοδήματος για όλους τους πολίτες και υπάρχει αυτός ως πρωτοβουλία πολιτών. Ε, πρότειναν να ενισχυθεί η οικονομία της γνώσης η οποία θα αντιμετωπίσει τις μελλοντικές οικονομικές προκλήσεις. Και όλα αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε την τελική έκθεση όπου περιλαμβάνονται όλες αυτές οι στάσεις. Εν κατακλείδη, θέλω να αναφέρω ότι η διαδικασία G1000 δεν επηρέασε μόνο την κατάσταση στο Βέλγιο αλλά και διεθνώς. Στο Ρότερνταμ υπήρχε μια πρωτοβουλία πολιτών ε, για την ε, αστική ανάπλαση. Στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία υπάρχουν πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίες ε, έχουν δημιουργήσει προσπάθειες για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και πολλές στο πόλη στο Βέλγιο έχουν χρησιμοποιήσει τη δική μας πρωτοβουλία ως πρότυπο για τις τοπικές πρωτοβουλίες συμμετοχής. Ε, με δύο λόγια πρέπει να πούμε ότι η δημοκρατία των πολιτών είναι ολοζώντανη και η χρονιά αυτή, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, έφτασε την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να πω εδώ, όπως και πολλοί άλλοι που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ευθύνη, ότι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά τους πολίτες και να γίνει μια προσπάθεια να ξαναδημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των βάθρων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρωτοβουλία G1000 και τώρα ας δούμε τις ερωτήσεις. Έχουμε ουσιαστικά 11, 11 λεπτά μόνο, αλλά μπορούμε ίσως να συνεχίσουμε λίγο για να δούμε τώρα ε, τις ερωτήσεις. Γκούντι Γκούντεσμαν, παρακολουθείς όλα τα tweet που έρχονται αν έρχουν, έρθει σχόλια από τις 30 πόλεις που είναι συνδεδεμένες με την εκδήλωση αυτή και μέσω των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, να μας τα πεις. Πες μας τι σου λένε τώρα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη. Είμαστε γνώμονες. πολλά σχόλια και πολλές ερωτήσεις. Κάποιες γενικότερες ερωτήσεις για την κυρία Τουιράν και άλλους ομιλητές. Παραδείγματο χάρη, το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πορτογαλία. Λέει ότι τα αντιευρωπαϊκά κόμματα ε, αυξάνουν τη δύναμή τους. Μήπως αυτό θα σκοτώσει την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Υπάρχουν νομικά ε, ε, επιχειρήματα για να δούμε αν οι αρμοδιότητες είναι εθνική ή ευρωπαϊκή. Αυτό έρχεται από τη Λετωνία. Πολλές ερωτήσεις προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Παραδείγματος χάρη από το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πράγα. Τι μπορεί να κάνει διαμεσολαβητής για να διαμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γραφείο ε, Κοινοβουλίου των κάτω χωρών θα ήθελε να μάθει τι μπορεί να κάνει ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής που δεν μπορεί να το κάνει ο Ολλανδός διαμεσολαβητής. Ποια είναι η διαφορά το, από την Ισπανία θέλουν να γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος σας στη, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, κάτι που αναφέρθηκε, και επίσης ε, υπάρχει ενδιαφέρον για την εκλογή του νέου διαμεσολαβητή που πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες και θέλουν να ακούσουν ποια κατά τη γνώμη σας, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το κατάλληλο προφίλ του νέου διαμεσολαβητή. Η κυρία Ρέντινγκ αναχώρησε κρίμα γιατί υπάρχουν ενδιαφέρουσε ερωτήσεις που απευθύνονται και σε αυτήν που ενδεχομένως όμως θα μπορούσαν να απαντήσουν οι υπόλοιποι. Οι πολίτες λένε ότι δεν έχουν επιρροή. Το πιστεύετε αυτό ή απλώς δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό. Σας τα αφήνω. Γκούντι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, θέλω να πω στο, ακροατήριο, υπάρχει μία ερώτηση στην οποία μπορούμε απε, απευθείας να προχωρήσουμε. Ε, α, ο κύριος εδώ, η πρώτη ερώτηση. Καλημέρα σε όλους. Ε, Ιταλός είμαι. Μάριο Ακάρντι το όνομά μου. Ήμουν διαμοσαλαβητής πριν από δέκα χρόνια στο Δήμο μου στη Σικελία, στο Καμπομπέλο Ντιμαντζάρα, στην επαρχία Τράπανη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διαμεσολαβητή για αυτή την πρόσκληση, γιατί έτσι μπορώ να συνεχίζω να ελπίζω σε αυτή τη διαμεσολάβηση. Ξέρει πολύ καλά ο διαμεσολαβητής τι θέλω να πω, γιατί το 2008 όταν ήρθε στο Παλέρμο το είχα πει και ανοιχτά δημόσια τότε ότι δυστυχώς στην Ιταλία, στην ε, Σικελία έχει πεθάνει η διαμεσολάβηση. Η δυνατότητα που έχουν οι πολίτες Δηλαδή κάποιος να τους ε, πάρει από το χέρι και να τους βοηθήσει να ακούσει τη φωνή σου. Δεν υπάρχει πια πέρα από τον διαμεσολαβητή που γνωρίζω τις δραστηριότητες του, τις ενέργειες του, θα ήθελα στην κυρία Ντουρά να ρωτήσω το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έκανε και επίσης τι ελπίζει να κάνει στο άμεσο μέλλον, ελπίζω να επανεκλεγείτε, ώστε να αποφύγετε να χάσουν αυτή την εμπιστοσύνη οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, αλλά η κύρια ευθύνη είναι των πολιτικών που έβγαλαν από τη μέση εκείνους που έπρεπε να υπερασπίσουν. Είναι ανόητο αυτό, ενώ αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να προσφέρουν μια υπηρεσία, να υπάρξει και ελπίδα επανεκλογής ε, και να αποφύγουμε την φωνή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρακαλώ. παρακαλώ. Καλημέρα σας, Στέλλα Βελική. Φυσικός ε, και σε θέματα πληροφορικής αρμόδια από την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Να συγχαρώ το Προεδρείο και την υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή γιατί από τότε που έμαθα την ύπαρξή τους σίγουρα διατήρησαν την ίδια επάρκεια ταχύτητα, αποτελεσματικότητα. Είναι ο μόνος θεσμός ίσως που ε, έχει μια άμεση επαφή σχέση με το Ευρωπαίο πολίτη. Ένα ερώτημα τώρα στους Έλληνες, στους Κύπριους, Ισπανούς, πώς θα τους ζητήσετε να συμμετάσχουν ε, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα πρέπει να τους εξηγήσετε τα προβλήματα που προκάλεσε η Τρόικα, τα λάθη τους, ε, τα λάθη της μεθόδου της Τρόικα. Και έτσι ίσως θα υπάρχει μια ευκαιρία να δείξουν ενδιαφέρον για σας. Και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη δεν πρόβλεπε όμως άλλες δυνατότητες. Για ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι πολίτες κάτι μπορούν να κάνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Άλλη μια ερώτηση αν μπορούμε να έχουμε. Ο κύριος Πίερς. Price. David το Έχω ένα ιστότοπο για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Ρέντινγκ. Πολλοί πολίτες ε, εξεπλάγησαν γιατί είδαν ότι η Κομισιόν προτείνει ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, πολιτικά δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν στη δημοκρατία, αποσύρεται το δικαίωμα δηλαδή όλων των πολιτών να είναι υποψήφοι για επίτροπη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ίσχυε από τότε που έγινε ο Ζωά Μονέ πρόεδρος. Δεν ήταν πολιτικός. Και άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν πολιτικοί. Με συγχωρείτε, μιλάμε για την οικονομική κρίση, κύριε Πράσι. Μιλάμε για την οικονομική κρίση. Νομίζω, νόμιζα ότι μιλάγαμε για τα δικαιώματα των πολιτών. Έχετε κάποια ερώτηση για την οικονομική κρίση, λέει ο πρόεδρο. Η οικονομική κρίση όμω ε, εξελίσσεται παράλληλα με την ε, ε, αποκλειστική χειραγώγηση των θεσμικών οργάνων από τους πολιτικούς. Πώς θεωρούν τα μέλη των, που είναι γύρω σα ότι θα ήταν δυνατόν να έχουν πάλι ε, όλοι οι πολίτε το δικαίωμα να γίνουν επίτροποι θα μπορούσαν να είναι όπω ο Χάλσταϊν ε, δικηγόροι, θα μπορούσε να είναι δημόσιοι πάλι, οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι μέλη τη Επιτροπή Πρόεδρο. Δεν έχουμε χρόνο για αυτή τη συζήτηση, αλλά να ακούσουμε τη Μαντάμ Ντουράν που ούτως άλλως θα πρέπει να φύγει. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ή να δώσω κάποια στοιχεία απάντηση σε αυτές τις παρατηρήσεις και στις ερωτήσει που ακούσαμε και από μακριά αλλά και από την αίθουσα αυτή. Για να δούμε πώς θα αποφύγουμε αυτό το αντιευρωπαϊκό αίσθημα που αναπτύσσεται να θανατώσει την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και μετά από αυτά που ακούσαμε για την κυρία ακριβώ για την εμπιστοσύνη, για την Τρόικα. Γιατί η Τρόικα θα πρέπει να αιτιολογήσει τις ενεργές της και να πει ότι εντάξει θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα λάθη, να αναγνωρίσει τα λάθη ενδεχόμενα και οι υποψήφοι για τις εκλογές, ίσως όχι για την Προεδρία της Επιτροπής γιατί δεν εκλέγεται άμεσα, δεν εκλέγονται άμεσα, αλλά να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα λάθη τους ή τουλάχιστον εκεί που έχω την εντύπωση ότι δεν βοήθησαν αυτή την δινή οικονομική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν αρκετοί από την Νότια Ευρώπη. Και εγώ, κυρία μου, δεν σας το κρύβω ότι ανησυχώ επίσης για την ψηφοφορία, όχι μόνο για τη συμμετοχή, αλλά και για την ψήφο που θα εκφράσουν οι πολίτες αυτές που θεωρούν τον εαυτό τους εντελώς να έχει εγκαταλειφθεί. Εντάξει, πέρα από αυτό, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος ε, είναι συνυπεύθυνος κλπ. Αλλά η Ευρώπη λένε ότι γενικά, γενικά, είναι υπεύθυνο έτσι χωρίς όνομα αλλά γενικά και θα πρέπει και να εξηγήσουμε όχι μόνο μας αυτό γιατί ακριβώς ε, είμαστε αφιψηλού και λέμε εγώ κατάλαβα θα σε εξηγήσω το τι συμβαίνει και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ακούσουμε, να αφήσουμε να εκφραστεί η οργή για να γνωριστούν τα λάθη αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διαφορετικά θα σε ακούσει κανείς τώρα σε αυτές τις χώρες. Αν δεν πείτε ότι έχουν ήδη διαπραχθεί λάθη, τότε δεν θα σας ακούει κανείς πια. Και ακόμα κάτι θεωρώ ότι το θέμα όπως είπα πριν είναι να δείξουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ναι, αυτό το δημοσιοέλλημα θα πρέπει να το ε, λύσουμε το θέμα αυτό. Διαφορετικά δεν θα έχουμε καμιά πολιτική, αλλά οι μέθοδοι ίσως δεν είναι και καλές. Ε, θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα και μετά να επιτρέψουμε να εκφράσουν την οργή τους, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και τέταρτο υπάρχουν και άλλες ε, αξίες εκτός από τις οικονομικές. Εντάξει, με λόγω της κρίσης δεν υπάρχει πια δυνατότητα περιθώριο για να μιλήσει κανείς για τίποτα, αλλά αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η πραγματικότητα η καθημερινή για πάρα πολλούς πολίτες. Φοβόσαστε όπως και από την πορτογαλική πλευρά τι ότι μπορεί να θίξει αυτό, τι, να σκοτώσει, να θανατώσει την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ναι, σίγουρα απάντηση. Και την εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ηθαγένεια η δυνατότητα. Νομικά υπάρχει το δικαίωμα ψήφου, διάφορα άλλα ευρωπαϊκής φύσεως δικαιώματα, αλλά επίσης και το πώς αισθάνεται κανείς από ευρωπαϊκής πλευράς. Αυτό είναι σε κρίση λόγω της κρίσης, έστω και αν δεν είναι υπεύθυνη για τα πάντα η Ευρώπη, έτσι όμως τη θεωρούν και ακόμα και το ευρωπαϊκό σχέδιο ορισμένο. Η ίδια η Ευρώπη αφισβητείται και η άκρα δεξιά εκεί που λένε ότι αλλά και από την ακραριστερά ε, πολλές φορές η ακραίοι είναι υπέρ μιας επαναδικοποίησης πολιτικής γιατί έτσι αυτός ο τρόπος όλοι μαζί να ενεργούμε δεν λειτουργεί και αυτό σύμφωνα και με την κλίμακα αρμοδιοτήτων όπως είπε κάποιος ναι ε, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση του κόσμου εντάξει δεν θα πρέπει ακριβώς να ξέρει ο πολίτης ποιος έχει ποια αρμοδιότητα, αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι τα διάφορα επίπεδα επικοινωνούν, συνομιλούν, συντονίζονται για να δώσουν συντονισμένες απαντήσεις ανάμεσα στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν το πιστεύει αυτό, γιατί ο καθένας στέλνει τον μπαλάκι στην απέναντι πλευρά, δεν φταίω εγώ, φταίω απέναντι. Η Αλεσάνδρα ίσως θα μπορούσε να μας πει μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Έχω την ερώτηση για τη σχέση του διαμεσολαβητή με τους πολίτες και τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Πεστε μου παρακαλώ, πώς κινητοποιήσατε τους ε, συμπολίτες σας για να υπάρξει αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Συνεργαστήκατε με τον ε, διαμεσολαβητή επ' αυτού. Η κυρία Μιράμπηλε. όχι δεν συνεργαστήκαμε συγκεκριμένα πρακτικά με τον διαμεσολαβητή για να κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, για να τους συνειδητοποιήσουμε να τους ενημερώσουμε για την εκστρατεία μας, όχι κατευθείαν με τον διαμεσολαβητή, αλλά συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. διότι μας υποστηρίζουν περίπου 50 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ένα βαθμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμαστε, ούτω ώστε να ενημερώσουμε για την ύπαρξή μας και δουλεύουμε επίσης και στα κοινωνικά μέσα πάρα πολύ, Facebook, Twitter, όλα τα κοινωνικά μέσα. Βέβαια δεν αρκεί αυτό, δεν αρκεί μόνο ε, να ε, είμαστε μέσα στα κοινωνικά μέσα. Πρέπει να έρθει κανείς και σε προσωπική επαφή με τους συνανθρώπους του για να τους ενημερώσει για όλα όσα κάνουμε. Για αυτά που είπε η κυρία Γκούτμαν ότι οι πολίτες έχουν την ε, αίσθηση ότι δεν μπορούν να παρέμουν βέβαια, βεβαίως έχετε δίκιο, αυτό οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα των θεσμικών οργάνων, πάντα υπάρχει κοινή ευθύνη. Επίσης και οι πολίτες θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο, να είναι πιο ενεργοί, να αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες, να προσπαθούν να βρουν την πληροφόρηση, να καταλάβουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, τι δυνατότητες έχουν να επηρεάσουν την ε, ενωσιακή νομοθεσία, τουλάχιστον να εκφραστούν επ' αυτής. Πρόεδρος, ε, σύντομα ο Ντιδιέ, κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ε, έχουν να κάνουν τι ρόλο μπορεί να παίξει ο διαμεσολαβητής, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, τι ρόλο μπορεί να παίξει το επίπεδο βάσης. Γιατί διαλέξατε το επίπεδο βάσης, το τοπικό επίπεδο και όχι τις άλλες δυνατότητες. Ε, το ευρωπαϊκό σύστημα είναι εξαιρετικά ελιτίστικο και θεωρήσαμε ότι μια πρωτοβουλία από τη βάση θεωρήσαμε ότι θα δώσει θα έχει την πρωτοβουλία και θα καταφέρει να ξεμπλοκάρει το σύστημα, να ξεπεράσει το αδιέξοδο. Είμαι όμως πιο θετικός όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης πάνω στους πολίτες. Πιο θετικά τα βλέπω από την κυρία Ντουιράν. Επί της ουσίας, σε πολλές χώρες, Ιρλανδία, Ιρλανδία ας πούμε, έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση τα τελευταία χρόνια και αυτή τη στιγμή οργανώνει μια συντακτική συνέλευση όπου ε, οι πολιτικοί και οι απλοί πολίτες συζητούν για το πώς θα μπορέσουν να οργανώσουν ε, δημοψήφισμα. Η Ισλανδία, το ίδιο, μια πολύ ε, δυνατή πολιτική, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και βλέπουμε ότι οργανώνεται φόρουμ πολιτών για να ξεμπλοκάρει το σύστημα να το κάνει καλύτερο. Και στο Βέλγιο είχαμε μια μεγάλη πολιτική κρίση, βαθύτατη, και διαπιστώσαμε ότι η κρίση αυτή αποτέλεσε πρωτοβουλία για ε, συζήτηση να σηκωθούν οι πολίτες για να αναλάβουν τον έλεγχο, να δείξουν ότι οι διαφορές μπορούν να ξεπεραστούν. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει πολιτική προθυμία. Αυτό γίνεται σε πολύ σε βάση των πολιτών για να δείξουμε ότι δεν εξαρτώμαστε από τα πολιτικά κόμματα, ότι δεν εξαρτώμαστε από την δημόσια χρηματοδότηση, εξαρτώμαστε από τους πολίτες και ότι οι πολίτες μπορεί να κινητοποιηθούν για να συμμετάσχουν ακόμα και χωρίς μια ε, επίσημη δομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντιντιέ. Να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ μερικές φορές ε, μέσω των κρίσεων υπάρχουν δεσμεύσεις ή ικανότητες από τους πολίτες για εναλλακτικέ λύσεις αλλά είμαι σε άλλη φάση εγώ στο τέλος τέλος πάντων ε, στη διαδικασία. Αυτή η κατάσταση έρχεται στους πολιτικούς, δηλαδή κάνει πηγαίνει δηλαδή σαν σέρ... Εδώ εντάξει δεν έχω αρνητική στάση, έχω τεράστια διάθεση, πολύ ενθουσιασμό στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας που θα ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι ο δυναμικός χαρακτήρας για μια δέσμευση είναι τέτοιος που ίσως μερικές φορές υπάρξει και υποδοχή κατάλληλη από του πολιτικού διαφορετικά θα μας απογοητεύσει η συμμετοχή ακόμα και στο Σύνταγμα το Ισλανδικό ή στην Ιρλανδία. Τώρα τα άλλο ίσως δημιουργήσουν νέες, ε, νέες καταστάσεις, ε, πράγματα νέα που θα μπουν μέσα στο Σύνταγμα που θα τα προκαλέσουν οι πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν που ίσως δημιουργήσουν προβλήματα και οι, ε, οι Βέλγοι πολιτικοί δεν τα υποδέχτηκαν με διαταδεσμό πολύ, είπαν α όχι όλα αυτά τα πράγματα παλιότερα ήταν φλιαρία, σε τίποτα και μεταξύ ε, σχημάτισα μια κυβέρνηση, αλλά μεταξύ τα πράγματα δεν είχαν να κάνουν ακριβώς με τη σύνθεση της όλης κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πριν αναχωρήσει η κυρία Ντιράν, να προσθέσω κάτι. Εμείς ε, στο γη χίλια. Ε, Λάμπρε Κριστίνα εκπρόσωπος του Βελγίου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το χωρίς περιορισμούς ε, βασικό εισόδημα. Ναι, για τους πολιτικούς, για τους πολίτες ε, θα πρέπει να υπάρχει μια επαφή. Πώς το βλέπω εγώ. Εδώ χρησιμοποιείται ένα μέσο που μας έδωσε η Ευρώπη αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αλλά εγώ είμαι μια απλή μεμονωμένη πολίτης και είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε επαφή με τους πολιτικούς γύρω από μένα γιατί μου κλείνουν την πόρτα, ασχολούνται πάντα με κάτι πιο ενδιαφέρον από το δικό μου και πρόκειται για μια επιτόπου μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Αρκετοί πολίτες να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και να έχει έτσι κανείς τη μικρή, την ισχνή ελπίδα και ελπίζω να μας ακούσει, να μας ακούσει μετά επιτέλους οι ε, πολιτικοί να ε, βρίσκουν τα αυτιά τους και να πούνε αυτή είναι πρωτοβουλία των πολιτών, θα πρέπει να την δούμε, να την εξετάσουμε γιατί έτσι οικοδομείται η Ευρώπη. Συμφωνείτε, ναι, συμφωνώ και ελπίζω ότι σε αυτή την πρωτοβουλία και καλή τύχη σε εσά να πετύχει, αλλά όπως είμαι και εδώ από την Επιτροπή Αναφορών που ιδιαίτερα έχει δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό, όταν ακριβώς όλα αυτά θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν πει όχι, έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον να υπάρξει μια συζήτηση. Αυτά που είπατε να εξεταστούν εκεί και όσα δεν μπήκαν από το παραθυράκι της Επιτροπής να μπουν από την πόρτα του Κοινοβουλίου για να συνεχιστεί όλη η συζήτηση. Και μια κάποια στιγμή αυτή η πρωτοβουλία σας να θριαμβεύσει. Αυτή είναι η δυνατότητα για να δοθεί μια συνέχεια σε αυτήν την εργασία σας ε, για να μην ε, ε, σταματήσει μόνο και μόνο επειδή θα πει όχι η Επιτροπή. Άρα λοιπόν οι πόρτες είναι ανοιχτές, λίγο λίγο σπρώξτε Ναι, θα αλλάξουμε τώρα τη σύνθεση των ε, ομιλητών μας. Εδώ μετέχουν. Ευχαριστούμε την Ασάντρα Μιράμπλε, Μάρκ Μπερτράν και Διδιέ Καλβέρτς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρέπει να φύγει η Ζαμπέλ, οπότε παρακαλώ ευχαριστήστε τους προηγούμενους ομιλητές. And in the meantime, we're going to... Εν τω μεταξύ θα καλέσουμε το δεύτερο πάνελ που περιλαμβάνει τον Επίτροπο Τσέρκοβιτς, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο για τις διαθεσμικές σχέσεις και την διοίκηση. Καθώς ε, χαιρετούνται οι ομιλητές, ο κύριος Σάρκοβιτς θα μας κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Δυστυχώς δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Ε, ο συναγερμός για τη φωτιά μας ε, το εξήγκλησε το διάλειμμα και επειδή ο χρόνος περνάει, θα προχωρήσουμε κατευθείαν στα σχόλια του Επιτρόπου. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρνς, ε, κύριε Διαμεσολαβητά, Νικηφόρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος πρότεινε αλλά και ε, οργάνωσε, είναι ο οικοδεσπότης αυτής της εκδήλωσης. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κατέβαλε προσωπικά, αλλά και το γραφείο του, οι συνεργάτες του, για να δείξουν πραγματικά πώς το γραφείο του διαμεσολαβητή μπορεί να προσεγγίσει τους πολίτες και να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες ε, ε, αισθάνονται ότι όταν υποβάλλουν ε, μια καταγγελία κάποιος θα την αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και θα προτείνει λύσεις. Στην ε, καριέρα του και λόγω της πολύ μεγάλης δραστηριότητας του γραφείου του το γραφείο του έδωσε μια φωνή στους πολίτες και υπερασπίστηκε τα συμφέροντά τους όταν χρειάστηκε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί την ε, εκδήλωση αυτή να τους ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχα με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου σε κάθε προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, να μπει αυτή στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω επίσης να επισημάνω την ε, στενή συνεργασία μας με την Επιτροπή Αναφορών, η οποία τα τελευταία χρόνια και λόγω της στενής σχέσης της με τους πολίτες έχει αποκτήσει εμπιστοσύνη και συνεργάζεται στενά με τους πολίτες και βεβαίως ε, κρατά σε εγρήγορση, δίνει πολλή δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτή είναι η Επιτροπή που αποφασίζει ποια είναι η αναφορά που θα, πάνω στην οποία θα δουλέψει και θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πια όχι. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Αναφορών, αλλά κυρίως τον διαμεσολαβητή για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Τώρα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε το νέο εργαλείο, το νέο μέσο, πώς τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών μπορούν ε, να έρθουν σε επαφή πιο αποτελεσματικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πώς ε, θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσεγγίσει τους πολίτες. Ξέρω ότι ακούσατε την κυρία Ρέντινγκ, τη συναδελφό μου σήμερα το πρωί, η οποία λεπτομερέστατα σας περιέγραψε την κατάσταση. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το έτος 2013 που είναι Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών για να προσεγγίσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από πλευράς θεσμικών οργάνων, τους πολίτες. Να λάβουμε υπόψη μας τη συλλογική σοφία των Ευρωπαίων πολιτών για το τι μπορεί να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια, να δημιουργηθεί μια ευκαιρία ε, αλληλεπίδρασης. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά φέτος για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες χρησιμοποιούν το νέο αυτό μέσο να επηρεάσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και για πρώτη φορά διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα ε, ολοκληρώσει τον πρώτο της πλήρη κύκλο. Με κάθε σεβασμό πρέπει να πω ότι τα, την αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά. Είναι η πρώτη ε, υπερεθνική συμμετοχική δημοκρατία αυτή, ένα εργαλείο για αυτού του είδους τη δημοκρατία. Την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και σοβαρότητα. Τι εννοώ. Διαπίστωσα ότι από τότε που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, έχουμε λάβει 25 αιτήματα εγγραφής τέτοιων πρωτοβουλειών. Τα, οι 14 έχουν ήδη εγγραφεί και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται πρωτοβουλίες για να φτάσουν το όριο του 1 εκατομμυρίου υποστηρικτών. Και αν επιτευχθεί η απαραίτητη γεωγραφική ισορροπία, τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη, θα περάσουν στην επόμενη φάση. Την επαλήθευση των υπογραφών από τα κράτη-μέλη, ακρόαση στο Κοινοβούλιο και κατόπιν συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν η Ευρωπαϊκή δηλαδή πρωτοβουλία μπορεί να γίνει ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε εκπροσώπους εδώ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών Πολιτών που παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους, έχουν περάσει αυτό το όριο έχουν το δικαίωμα να κάνουν ε, αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν ξεπεράσει τα ε, ένα εκατομμύριο μέλη και ε, πλησιάζουν στην, επιτυχή, στην επίτευξη αυτής της γεωγραφικής ισορροπίας. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε για αυτές τις εμπειρίες θετικές και αρνητικές συγκέντρωσης υπογραφών. Ακούσατε, και δεν θα το κρύψω, ότι υπάρχουν, υπήρξαν κάποια προβλήματα κάποιες παιδικές ασθένειες ε, που έχουν σχέση με τα ε, διαδικτυακά συστήματα συγκέντρωσης ε, υπογραφών, όπως επίσης και της αναγνώρισης και της εισαγωγής. Όλα αυτά ήταν αναμενόμενα, γιατί αν ξεκινά κανείς μια προσπάθεια τέτοιου εύρους όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πρέπει να, έχει, να ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να δείξει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, να βοηθήσει όσο μπορούσε την εγκατάσταση του λογισμικού open source να προσφέρει δυνατότητα από το Λουξεμβούργο να βοηθηθούν οι οργανωτές και να ε, πιστοποιηθούν από τις αρχές του Λουξεμβούργου οι οργανωτές. Πρέπει να πω πολλά καλά για τις γερμανικές αρχές που κατάφεραν να εισάγουν τις διαδικασίες επαλήθευσης με υποδειγματικό τρόπο. Το δικαίωμα ε, στην πρωτοβουλία αυτή για το νερό στηρίζεται στην γερμανική προσέγγιση. Δείχνει ότι όταν υπάρχει καλή διοικητική προσέγγιση και πολιτική θέληση όλα αυτά είναι εφικτά. Και αυτό θα εξυπηρετήσει και τους κατοίκους του Λουξεμβούργου και της Γερμανίας και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Πολύ σημαντικό είναι ότι οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών συνεισφέρουν στο να ξεκινήσει αυτό που εγώ αποκαλώ μια πραγματικά πανευρωπαϊκή συζήτηση μεταξύ πολιτών. Είδαμε το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών μέσων που διευκόλυναν πάρα πολύ την αλληλεπίδραση αυτή πέρα από τα σύνορα και επέτρεψαν στους Ευρωπαίους πολίτες να διατυπώσουν σκέψεις, ανησυχίες, φόβους και ελπίδες και ιδανικά. Όλα αυτά θεωρώ ότι αποτελούν ένα μόνο πρώτο βήμα για αυτό το οποίο θα δούμε στο μέλλον. Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία υπερεθνικής ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοκρατίας. Τώρα υπάρχει η η πληροφορική, η πιστοποίηση, η επαλήθευση, όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Όπως θα υπάρχουν οι ε, ηλεκτρονικές ταυτότητες και οι άλλες ηλεκτρονικές δυνατότητες, πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα τις χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο αν είναι πολύ πιο φιλικές στο χρήστη μορφές τους. Δεν θα χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες μόνο για την ε, αποθήκευση των ιατρικών και άλλων δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν και ε, σε ε, συζητήσεις αλλά και στις εκλογές όπως είδαμε ότι γίνεται στην Εσθονία. Και έτσι θα υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα για τους πολίτες να, με ένα κλικ να είναι δίπλα σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές συζητήσεις. Θα αποκτήσουν πολύ ισχυρότερη θέση στην δημοκρατία της Ευρώπης σε λίγα χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί προς την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Όταν θα αποκτήσει η Επιτροπή ε, νέες δυνατότητες για τους προϋπολογισμούς ή για να κάνει συστάσεις για θέματα ε, φροντίδας των παιδιών κλπ. που στο παρελθόν θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό εσωτερικά ζητήματα. Ταυτόχρονα είναι προφανές ότι θα ζητήσουν οι πολίτες όλο και περισσότερο ε, αυτή, η δημοκρατική διαδικασία να ενισχυθεί, να ακούγεται η φωνή τους, να συμμετέχουν στις συζητήσεις που αφορά την στενότερη οικονομική συνεργασία. Θα δούμε λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια υπερεθνική δημοκρατική διαδικασία για τη συζήτηση αυτή, η νέα γενιά του Facebook και του Twitter θα χρησιμοποιήσει τα μέσα της συμμετοχικής δημοκρατίας όπως τις πρωτοβουλίες πολιτών, όλο και περισσότερο στο μέλλον. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι χάρη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών οι πολίτες έχουν μια πραγματική ευκαιρία να εκφράσουν τις ελπίδες, τις απόψεις και τις ανησυχίες τους με τρόπο πιο συγκεκριμένο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ακούγονται στα θέματα η φωνή τους και να συζητείτε στην Ευρώπη αυτό το οποίο επιθυμούν. Έχει γίνει ακριβώς αυτό. Η, πρώτη, η αδερφότητα 2020 ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που καταγράφηκε και όπως είπα βρίσκεται ακριβώς το πριν την ολοκλήρωσή της, πριν φτάσει στο απαραίτητο όριο όχι μόνο του συνολικού αριθμού υπογραφών, αλλά και της απαραίτητης γεωγραφικής κάλυψης, ώστε να θεωρείται ότι δικαιούται αυτή η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ότι έχει καλύψει όλο το πεδίο για να περάσει στη δεύτερη φάση. Αν δούμε τώρα και αυτή αλλά και πολλές άλλες πρωτοβουλίες πολιτών διαπιστώνουμε ότι αποκρίνονται πραγματικά στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες για τα θεμελιώδη ωφέλη και δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα ευρέ, ε, γνωστά θέματα, αλλά και θέματα που για διάφορους λόγους έχουν ξεφύγει από την προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και υγιές για τις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουν οι πολίτες να ακούγεται τη φωνή τους σε θέματα ζωής, δουλειάς, να πούν πράγματα που αφορούν την υγεία, ε, να μιλήσουν για τους πολίτες και για τον πλανήτη. Θέλουν να ζουν σε μια κοινωνία όπου θα είναι σεβαστή η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που καλύπτουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών και θα δούμε πολύ περισσότερα όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος με επιτυχία. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη επιθυμία να συναντηθούν οι οργανωτές και γι' αυτό ήταν καλό που μπήκε η ρήτρα θεώρησε στο πρώτο κύκλο, γιατί πιστεύουμε ότι θα μάθουμε πολλά από αυτόν τον κύκλο. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει, πιστεύω, να κάνουμε ακόμα πιο φιλική στους χρήστες την όλη αυτή διαδικασία και πραγματικά πιστεύω στο μέλλον των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών των Πολιτών που θα μπορέσουν να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες που θα ε, αντιδρούν πολύ πιο άμεσα ώστε οι πολίτες ε, να αισθάνονται ότι πραγματικά αν κάτι τους απασχολεί πολύ, αν θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, υπάρχει ο τρόπος να γίνει αυτό. Είναι η στιγμή που πρέπει το μέσο αυτό να το καλλιεργήσουμε, να το διευρύνουμε και να το κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικό στους χρήστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε Σεφκόιτς. Και τώρα να παρουσιάσω τα μέλη που είναι εδώ γύρω μου, που έχουν αλλάξει από προηγουμένω. Πρώτα απ' όλα εδώ, δεξιά του κυρίου Σεφκόιτ, είναι ε, ο Πίτερ Γκέρτσε. Εδώ συζητάμε για το πώς πρέπει να απευθυνθεί κανείς στο διαμεσολαβητή και πώς θα σας βοηθήσει ο διαμεσολαβητής να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση, για παράδειγμα, διαφάνειας ε, ιατρικών δεδομένων για ε, φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εδώ, στο, στα δεξιά μου, στο, μέλος του, στο τέλος του τραπεζιού, είναι ο Κεροζάνερ Νόβακ, είναι επιχειρηματίας από την Εστονία, έχει μια σειρά από επιχειρήσεις ε, πληροφορικής, είναι επίσης επικεφαλής μέσα οργάνωση για τη φύση και είναι επικεφαλής και μέσω οργάνωση που λέγεται «Ας το επιχειρήσουμε» είναι μια οργάνωση βάσης που είναι από τις πιο ταχεία επεκτηνόμενες οργανώσεις πολιτών στην ιστορία που θέλει να κινητοποιήσει την Ευρώπη για να καθαρίσουμε το περιβάλλον. Και δίπλα στο Άινορ είναι η Αν Μαρή Περέ, είναι επικεφαλής της πρωτοβουλίας των πολιτών, της Επιτροπής Πολιτών που προωθεί μία αναφορά για να υπάρξει ε, καθαρό πόσιμο είδωρ και αποχέτευση στην Ευρώπη είναι πρωτοβουλία των πολιτών, έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφέ και στόχος είναι τα δύο εκατομμύρια είναι επιπλέον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία ε, Συνδικάτων Δημοσίων Υπαλλήλων. Θέλουν ε, βεβαίως να καταπολεμήσουν και την ιδιωτικοποίηση της αγοράς υδάτων στην ε, Ευρώπη. Έχουμε πολλές ερωτήσεις που λαμβάνουμε και από τα γραφεία του Κοινοβουλίου που συνδέονται με την εκδήλωσή μας ε, μέσω του streaming καθώς και μέσω των ε, tweets που λαμβάνουμε από ολόκληρο τον κόσμο. Όπως σας είπα το hashtag είναι EYC2013EO στα αγγλικά. Η Γκούντι βλέπω ε, του γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή βλέπω ότι παίρνει πολλά tweets τα οποία εισραίουν εδώ στο τείχος από tweet. Να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην Αν Μαρή Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρνα. Επίση, τον κύριο Διαμαντούρο, διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωση και όλοι συνεργάτες του. Ε, να ευχαριστώ, το καλώς ορίσατε. Καλημέρα σε όλους όσους είναι παρόντες, αλλά και όλους όσους μας βλέπουν ή τουλάχιστον μας ακούν από μακριά και που επίσης υποβάλλουν ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω και ε, βάση αυτής της ε, πρωτοβουλίας ε, στις ελευθερία λοιπόν, μας, τον Ζέρι Βαντεμπέργκ, γιατί είναι εκείνος που στους ώμους του φέρει κατά κύριο λόγο αυτή την πρωτοβουλία, τον Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Κύριε Σέσκοβιτς, σας ευχαριστούμε για τα λόγια σας ε, για θέματα της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, όπως το είπατε και ο κ. Κρις Μπέρν το υπενθύμησε. Σίγουρα περήφανοι είμαστε που ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο 360.000 άτομα, αλλά θα πρέπει να περάσουμε κι άλλη μια φάση, μια ισορροπία γεωγραφική ανάμεσα στις διάφορες χώρες και θα επανέλθω στο θέμα αυτό στην ε, Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία μαζί με άλλους, μαζί με μη κυβερνητικέ ευρωπαϊκές οργανώσεις. Εποφεληθήκαμε από το παγκόσμιο επίπεδο και σε, στον ΟΗΕ γιατί είναι η το Διεθνές Έτος Συνεργασίας για θέματα υδάτων και επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το έτος που είναι των Ευρωπαίων πολιτών. Για το είδωρ να υπενθυμίσουμε τα εξής. Το 2000 είχαμε μια οδηγία για το νερό και αναφέρεται ότι δεν είναι ένα εμπόρευμα, δεν είναι μια commodity, δεν είναι εμπορική υπηρεσία όπως ακριβώς ε, συνηθίζουμε να το παρατηρούμε για άλλα αγαθά τα οποία ενώ το νερό είναι ένα κοινό αγαθό και στο ΛΟΗ είχαμε αυτό το ψήφισμα το 2010 που μας επέτρεψε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε και που θεωρείται ότι το νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και πάνω σε αυτό κυρίως βασίσαμε την όλη εκστρατεία μας το δικαίωμα στο νερό. Και επίσης ε, στήκαμε στην συνθήκη της Λαβώνας ώστε μέσω αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών να πετύχουμε να ασχοληθεί σοβαρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νομοθεσία για το νερό διότι το νερό είναι κοινό αγαθό και δικαίωμα και όχι απλά ένα εμπόρευμα το οποίο έχει να κάνει με το συνολικό ανταγωνισμό. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα βρισκόμαστε εδώ και θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντούρο επιθυμούμε μέσω αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών εσείς ε, σαν Ευρωπαίοι πολίτες να δεχτείτε ενεργοί και μετά από μια σύντομη παρουσίαση πόντ κλπ. θα ήθελα να σας παροτρύνω να υπογράψετε και να προωθήσετε και σε άλλους για να υπογράψουν αυτή την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Παρακολουθώ τους τεχνικούς να ξεκινήσει η προβολή του βίντεο. En 2010, les Nations Unies reconnaissent le droit universel à l'eau et l'assainissement, essentiel à la réalisation de tous les droits de l'homme. Cette initiative était censée augmenter l'accès à l'eau et l'assainissement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 signer la pétition. Παρακαλώ, μήπως θα μπορούσε να ξεκινήσει και η παρουσίαση PowerPoint ε, για να δούμε στα γρήγορα πώς έχει κατάσταση, ναι είναι δικαίωμα των πολιτών. Χρειάζεται νερό για όλους. Αλλά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτός ο διτός χαρακτήρας, ένα δικαίωμα, πώς μπορεί κανείς να τον εντυπίσει σαν θεμελιώδες δικαίωμα και από την άλλη μεριά όμως ε, Εάν είμαστε στα πλαίσια μιας αγοράς και ενός ανταγωνισμού, αυτού που μας ζητούν καθαρά είναι ακριβώς να μην υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα, γιατί κατά την άποψή μας είναι δημόσιο αγαθό και πρόκειται για μια υπηρεσία ουσιαστική που έχει δημόσιο χαρακτήρα για όλους. Και τι έχουμε σαν απαιτήσει. Η προμήθεια σε νερό, η επεξεργασία του νερού να μην υπόκειται στους νόμους του ανταγωνισμού της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει σχετικά, να ρυθμίσει την κατάσταση για την πρόσβαση στο νερό και στα 27 κράτη-μέλη και για την κατάλληλη επεξεργασία του και ακριβώ όπως για, τον, ε, για το φόρο ντόμπινγκ ρομπέτων δασών, αυτά που ακριβώς που έγινε, υπόθηκαν από τον ΟΗΕ να αποτελέσουν πραγματικότητα, να υπάρχει παγκόσμια δυνατότητα πρόσβαση στο νερό με μια κατάλληλη επεξεργασία του για να μην είναι επικίνδυνο. Τι επιθυμούμε εμείς μέσω του 1.360.000 περίπου υπογραφών η όλη αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως έχω μια άμεση ερμηνεία της θέσης Επιτροπής ε, να υπάρξει μια κατάλληλη τοποθέτηση όχι όπως τώρα από την αγορά και τον αγωνισμό να κατευθυνθεί προς ε, μια θέση κάτι που έχει να κάνει με το δημόσιο αγαθό και σαν δικαίωμα μέσω αυτής της πρωτοβουλίας των Ευρωπολιτών το σημαντικό είναι ο κόσμος να έχει τα μέσα να ενεργήσει άμεσα και τι αντιληφθήκαμε ότι οι πολίτες, ε, για τους πολίτες τι τους απασχολεί το νερό που το αντιμετωπίζουν σαν δημόσιο αγαθό. Δεν θέλω να σας διαβάσω τώρα τα πάντα που συνοδεύουν αυτή τη διαφάνεια και επειδή είναι και στα γαλλικά, ας τα αφήσουμε λοιπόν, αλλά να υπενθυμίσουμε το πρόβλημα αυτό ανάμεσα σε θεμελιώδες βασικό δικαίωμα και πρόσβαση σε όλους. Και τον Απρίλιο που μας πέρασε από την Βεόλια κάποιος ε, απολύθηκε γιατί είχε αρνηθεί να διακόψει την παροχή νερού σε κάποιον που δεν είχε τα οικονομικά μέσα. Και η Βεόλια τον ε, απέλησε γιατί σε πολυεθνική εταιρεία, λέει ότι η οικογένεια αυτή, έστω και αν δεν είχε χρήματα, δεν πλήρωνε το λογαριασμό της. Θα έπρεπε να της διακοπεί η παροχή. Και ακριβώς, λοιπόν, θα πρέπει να δοθεί και μια μάχη σε εκείνους, απέναντι σε εκείνους να τους πούμε που λένε ότι είναι μια εμπορική παροχή, ένα εμπόρευμα πρόκειται και ο Γενικός Διευθυντικός της Νεστλέ είπε λυπάμαι, ακούστε, εάν δοθεί ειδικό χαρακτήρα στο νερό, εντάξει γιατί όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Με τον κύριο Κρίσπερν συνομιλήσαμε πριν από λίγο. Στη Γαλλία έχουμε μια διπλή αντιμετώπιση. Εγώ ίδια είμαι Γαλλίδα και πρόεδρος αυτής της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας πολίτων και πολύ καλά γνωρίζω ότι στη χώρα μου, τη Γαλλία, τουλάχιστον δύο ισχυρέ παλαιδόνε, δηλαδή η Δεβεσουέντ και η Εόλια, που ασκούν ηγετικό ρόλο. Ε, στη Γαλλία αλλά και αλλού μας υποστηρίζουν τοπικοί εκλεγμένοι και εθνικοί επίσης και βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί ακριβώς προχάμε στη σύσταση μιας οργάνωσης σύμφωνα με τα όσα μας ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της σχετικής πρωτοβουλίας πολίτων και πώς εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε με άλλες οργανώσεις, βλέπετε τα ονόματά τους και προχωράμε στη σύσταση μιας Επιτροπής Πολιτών με 33 μέλη και στη συνέχεια προχωράμε στη σύσταση ομάδων ε, περιφερειακών και επίσης υπάρχουν και οι λεγόμενοι πρέσβεις, ε, πώς να σας το πω τώρα, ε, λίγο πολύ γνωστοί στις χώρες μας ε, και έτσι μπορεί να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία και στη Γερμανία ας πούμε, ε, κάποιος που κάνει σκίτσα χιουμοριστικά. προχώρησε ακριβώς στην όλη πρωτοβουλία γιατί με τον τρόπο του πρόθεσε την όλη πρωτοβουλία και ακριβώς πετύχαμε τουλάχιστον στη Γερμανία το έστωνε εκατομμύρια. Όπως λέει και ο Ομπάμα, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Πού βρισκόμαστε τώρα, σε ποιο σημείο, σε αυτή την ισορροπία, αυτή την περίφημη ισορροπία που πρέπει να πετύχουμε σε εθνικό επίπεδο, γιατί 1.360.000 υπογραφές, υπέροχο είναι, Τώρα όμως θα πρέπει να ανταποκριθούμε και σε άλλη ανάγκη κριτηρίων μια ισορροπία γεωγραφική στις χώρες μας και στη Γαλλία. Έχουμε 11.000 ενώ απαιτούνται 55.500 τουλάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό το μήνυμα θα ήθελα να σας απευθύνω. Πηγαίνετε στο ίντερνετ το Right to Water, δικαίωμα για το νερό και υπογράψτε και παροτρύνετε και τους γνωστούς και φίλους σας να υπογράψουν και εκείνοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που μας αφιερώσετε. Ευχαριστούμε την Αν Μαρή Πέρε. Αυτό είναι το αίτημα λοιπόν. Δούμε τώρα πώς αρέσει να το αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να υπάρξει μια καθαρή και υγιής Ευρώπη. Τίθεται το θέμα της υγείας των πολιτών. Αυτό θα μας πει ο Πέιτερ Γκέρτσε. Είναι επικεφαλής του Βορείου Κέντρου Υγείας. Το 2007 απευθύνθηκε στο διαμεσολαβητή, πήγε στον Νικηφόρο και του είπε «Κοίταξε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μας δίνει πρόσβαση σε κλινικές μελέτες και δοκιμές για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Παρακαλώ. Πέστε μας περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρουμε πώς να αξιοποιήσουμε με ασφάλεια και να χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια τα φάρμακά μας στην ε, Ευρώπη και τις ΗΠΑ τα φάρμακα είναι το τρίτο αίτιο θανάτου μετά την ε, καρδιοπάθεια και τους ε, καρκίνους. Ο σημαντικός λόγος γι' αυτό είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία αποκρύπτει τα στοιχεία για τα τι παρενέργειε των φαρμάκων του. Ε, δημοσιεύουν μόνο τι μισέ κλινικέ δοκιμέ του και αυτό που δημοσιεύουν είναι πολύ συχνά με σοβαρό τρόπο παραπλανητικό. Τα φάρμακα κατά τη παχυσαρκία είναι επικίνδυνα και γι' αυτό το 2007 ζητήσαμε πρόσβαση σε μη δημοσιευμένε μελέτες που είχαν αποστείλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Φαρμακοβιομηχανίες για να πάρουν ε, ε, άδεια εμπορίας. Ο επικεφαλής του οργανισμού αυτού, Τόμα Λούγκρεν, δεν μα έδωσε πρόσβαση και γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε στον διαμεσολαβητή. Τα επιχειρήματα του Λούγκρεν ήταν τα εξή. Προστασία εμπορικών συμφερόντων, ότι δεν υπήρχε επιτακτικό δημόσιο συμφέρον ε, διοικητικό βάρος για να μας παράσχουν και ότι δεν θα είχαν καμία αξία αυτά τα στοιχεία ε, ε, εφόσον ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα είχε αφαιρέσει διάφορα τμήματά του. Απορρίψαμε αυτά τα επιχειρήματα και ο διαμεσολαβητή συμφώνησε μαζί μα. Επιθεώρησε τα έγγραφα στα γραφεία του οργανισμού αυτού και συνεπέρανε ότι δεν περιείχαν καθόλου εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία. Αλλά ο Οργανισμός Φαρμάκων αντιστάθηκε εντελώς στα επιχείρηματα αυτά, δεν μας έδωσε πρόσβαση. Μόνο όταν ο διαμεσολαβητής το 2010 κατηγόρησε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για κακοδίκηση σε μια ανακοίνωση τύπου, τότε μόνο άλλαξαν τη θέση του και μας έδωσαν πρόσβαση στα στοιχεία. Ο Τόμας Λούγκρεν έφυγε από τον οργανισμό αυτό μερικού μήνε μετά και ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου για την φαρμακομηχανία. Κάτι που απαγορεύεται σαφώς από τους ιστορικούς κανόνες του οργανισμού αυτού που προβλέπουν μια περίοδο απαγόρευσης απασχόλησης στον ίδιο τομέα για δύο χρόνια. Ο νέος διευθυντής του οργανισμού Γκίντο Ράζι έχει πολύ διαφορετική άποψη για τη διαφάνεια. Από τον Ιανουάριο 2014 στόχο του οργανισμού είναι να παρέχει δημόσια πρόσβαση όχι μόνο σε όλα τα όλες τις μελέτες και τις δοκιμές, αλλά και στα κατέργαστα δεδομένα που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ελέγχουν οι ίδιοι όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι τρομερή πρόοδος για τη δημοσία υγεία. Αλλά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί να το αποτρέψει. Δύο φαρμακοβιομηχανίες έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και αν επιτύχουν θα αποτρέψουν την ε, αποκάλυψη των ε, φαρμάκων. Εάν το επιτύχουν αυτό θα συνεχίσουμε να δολοφονούμε τους πολίτες μας, τεράστιο αριθμό συμπολιτών μας και ασθενών μας, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα φάρμακα που τους χορηγούμε. Αυτό είναι σκάνδαλο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να αναθεωρήσει την οδηγία για τις κλινικές δοκιμές προτείνει να μας χορηγηθεί πρόσβαση σε συνοψίσεις των κλινικών δοκιμών. Αλλά αυτό δεν είναι επαρκές οι συνοψίσει πολλέ φορέ είναι παραπλανητικέ. Θέλουμε πρόσβαση συνολικά σε όλε τι μελέτε, σε όλο το κείμενο των μελετών και στα κατέργαστα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία για αυτά που χορηγούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μία για όλου του άλλου. Επίση θα αποφεύγονται οι απάτε. Θα μπορούμε να ελέγξουμε τι έχει κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό θα ήταν τεράστια πρόοδο για τη δημόσια υγεία. Με αυτόν τον τρόπο θα ε, υπήρχε περισσότερη καινοτομία στον ε, τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Διότι αν μια φαρμακοβιομηχανία μπορεί να δει τι λάθη έχουν κάνει οι άλλες φαρμακοβιομηχανίες, γιατί μπορούν να δουν τα στοιχεία, τότε μπορούν να αποφύγουν να επαναλάβουν τα σφάλματα αυτά. Μην το ξανάτε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάτι θεμελιωδώς λάθος με τον τρόπο με τον οποίο θέτουμε τις προτεραιότητές μας στην ε, περίθαλψη. εάν για λόγους εμπορικούς ή για λόγους σταδιοδρομίας κάποιων σημαντικά στοιχεία δεν είναι προσβάσιμα. Στοιχεία που είναι σημαντικά για λογικές και σωστές αποφάσεις από τους ασθενείς, για τους, από, τους, ε, συγγνώμη, από τους ιατρούς, για τους ασθενείς τους. Δεν θέλουμε επίσης να ζούμε σε κοινωνίες όπου υπάρχει μία μόνο εκδοχή της αλήθειας. Δεν είναι τρόπος αυτός για να λειτουργεί η επιστήμη. Η επιστήμη θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί από άλλους και όχι από αυτούς που έχουν τρομερό εμπορικό συμφέρον να κρατούν μυστικά τα δεδομένα και να χειραγωγούν και να τροποποιούν τα δεδομένα που δημοσιεύουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό τον επόμενο μήνα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα ψηφίσουν για τις τροπολογίες, για την οδηγία, για τις κλινικές δοκιμές. Ελπίζω οι ευρωβουλευτές να ψηφίσουν για να υπάρχει πρόσβαση όχι μόνο στη συνόψηση. Διότι αν έχουμε πρόσβαση μόνο στη συνόψη, πολλέ μελέτε θα πηγαίνουν χαμένες και θα εξακολουθήσουμε να εκμεταλλευόμεθα τους ασθενείς για εμπορικούς λόγους, για λόγους ε, προώθησης της σταδιοδρομίας μας. Όπως το καθαρό νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα, έτσι είναι και τα αξιόπιστα στοιχεία από την ιατρική έρευνα. Είναι θεμελιώδη δικαίωμα. Μας αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πίτερ Κούτσε και περνάμε αμέσως στον Ράινερ Νόλβακ, ο οποίος προλίγου είπε ότι έχει οργανώσει μια παγκόσμια εκστρατεία καθαρισμού που έχει λοιπόν τη σκοπιά της οργάνωσης της βάσης. Είδαμε τις άλλες πλευρές, να δούμε και τη σκοπιά της οργάνωσης από τη βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι προέρχομαι από ένα μικρό νησί στην ακτές της Εστονίας που, μου για το, από το οποίο χρειάζομαι μια μέρα για να έρθω εδώ και σκεφτόμουν πάρα πολύ, είχα τη δυνατότητα να σκεφτώ. Υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν το Twitter εδώ. Σας παρακαλώ. Αυτοί που ε, ε, πραγματικά ενδιαφέρονται για την Ευρώπη και είναι διατεθειμένοι να μείνουν εκεί ε, τρεις ώρες για να ακούσουν τι κάνουμε και να, εμείς να τους χειροκροτήσουμε. Να τους χειροκροτήσουμε. Ευχαριστώ. Είδα σχόλια του τύπου είναι βαρετό, είναι πολύ μεγάλες οι ομιλίες. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Έχω ένα όνειρο, ένα μικρό όνειρο, που ξεκίνησε στην από την Ιστονία. Ήταν πολύ συνηθισμένο μετά τη Σοβιετική περίοδο να πετάει κανείς τα σκουπίδια του στην εξοχή. Τόσο πολύ που είχα φτάσει στο σημείο να θυμώνω κι εγώ και φίλοι μου. Και θεωρήσαμε ότι θα κάναμε μια τελευταία απελπισμένη προσπάθεια για να γίνει κάτι. Και υπάρχει ένα μικρό βίντεο το οποίο θα σας δείξω σε λίγο για όλα αυτά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το δείτε.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 The third step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. see ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja, ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval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 Μίλησα με τον κύριο Διαμαντούρο και με ρώτησε αν μπορούσα να βοηθήσω για να συμμετέχουν οι πολίτες, γιατί αυτό ακριβώς κάνουμε. Για μένα η συμμετοχή των πολιτών, η εμπλοκή τους, η δέσμευσή τους, ε, είναι σαν να λέμε πώς κάνουμε το, τη μαϊμού να πηδήξει. Οι άνθρωποι είναι δεσμευμένοι, ασχολούνται το θέμα είναι πώς θα ασχοληθούν οι πολιτικοί στην πραγματικότητα. Άκουσα στην προηγούμενη συζήτηση ότι θα πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν. Νομίζω ότι θα πρέπει οι πολιτικοί να καταλάβουν. Δεν θα πρέπει να χειροκροτάτε. Αυτό δεν ήταν ένα καλό σημείο. Αυτό με πηγαίνει προς τη σκέψη η οποία θα μας οδηγήσει στη συζήτηση που ε, οδηγεί στην Ευρώπη όπου όλοι είναι θυμωμένοι με τους υπολείπους. Αν θέλουμε να συμφωνήσουμε με τη μία πλευρά μόνο, τότε θα, θα καταλήξουμε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή την πολυτέλεια δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι καλό είναι κάτι που κάναμε εκεί. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα των σκουπιδιών και το κάναμε ωραίο, ευχάριστο, πλάκα. Δεν είμαστε κίνημα για το περιβάλλον. Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν μ' αρέσει το, το, να μ' αρέσει να καθαρίζω, μ' αρέσουν όμως τα καθαρά πράγματα. Μ' αρέσει η καθαριότητα. Ίσως να το κάνω μερικές άλλες φορές, αλλά όχι και πάρα πολύ. Πέρυσι συμμετείχαν 96 χώρες σε παγκόσμιο καθαρισμό. Αυτό με ξεπερνάει. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι τα σκουπίδια που μαζεύουμε εκεί από το έδαφος. Περισσότερα σκουπίδια μαζεύουμε μέσα από το μυαλό μας. Αυτό κάνουμε. Κάνουμε κοινωνική αλλαγή. Αυτό κάνουμε. Λέμε στους ανθρώπους ότι είναι καλό να κάνουμε τα πράγματα όλοι μαζί, να έχουμε κοινέ αξίες. Περί αυτού πρόκειται. Και το πολύ σημαντικό για τη, με την βάση των πολιτών είναι ότι μπορεί κανείς να παραμείνει αυθεντικός, πιστός τα πιστεύω του. Αν δει κανείς τις οντότητες όπως είναι οι επιχειρήσεις, εκεί υπάρχουν η ιεραρχία. Και αυτό είναι καλό για την παραγωγή κουτιών, πολλών κουτιών. Αν εμείς θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν ως μηχανήματα κατανάλωσης, εντάξει. Αλλά αν όμως σκεφτούμε πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μία δομή δικτύου. Και οι ιεραρχίες έχουν πολλά πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί εμείς μπορούμε να κινηθούμε πιο άμεσα και πιο γρήγορα. Και ακριβώς γι' αυτό δεν ψηφίζουν οι νέοι η ψηφοφορία είναι κάτι που ανήκει στο 19ο αιώνα. Πράγματι, οι πολιτικοί που εκφωνούν μακροσκελείς λόγους, αυτό είναι εποχής 19ο αιώνα. Πρέπει να πει στους ανθρώπους πώς να εμπλακούν και να το συζητήσει κανείς. Οι άνθρωποι εμπλέκονται, συμμετέχουν από τη στιγμή που καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει νόημα. Και αυτό το έχω δει σε πάρα πολλά μέρη. Όπως ε, ο καθαρισμός που κάναμε πέρυσι στο Κωσυφοπαίδιο. Ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκε εκδήλωση σε εθνικό επίπεδο που 35.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και δεν ζήτησαν την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκαναν μια οργάνωση μόνο τους, μια ομάδα από τη Βοσνία, όπου οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί δούλεψαν μαζί σε μια ομάδα για να καθαρίσουν τη χώρα. Αυτό, πιστεύω, είναι κάτι το νέο που συμβαίνει εδώ ή μάλλον κάτι παλιό που το ανακαλύπτουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσο μοιάζουμε όλοι μας στην ουσία. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού. Ε, προσπαθούμε να βρούμε κάτι το καθαρό, το αγνό και αυτό έχει χαθεί από την πολιτική εδώ και πολύ καιρό. Μπορεί να με κατηγορήσετε, να μου πείτε ότι είμαι ιδεαλιστής, αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνονται τα πράγματα. Ονειρεύεσαι κάτι που είναι σωστό. Για μένα τουλάχιστον το όραμα, το όνειρο ενός, κοινού, ενός καθαρού κόσμου με κινητοποιεί. Μπορώ να πάω το νησί μου, στην ακτή, ε, μετά από μια καταιγίδα που έχει φέρει σκουπίδια από τη Δανία, τη Γερμανία ή τη Σουηδία, να τα καθαρίσω γιατί πιστεύω ότι και κάποιοι άλλοι στις δικές του ακτές αυτό θα κάνουν και τελικά ο κόσμος θα καθαρίσει. Δεν είναι τόσο παλιά, πριν από χίλια χρόνια περίπου, μπορούμε να μπορούσαμε να πίνουμε νερό από το Σικουάνα. Γιατί να μην το κάνουμε. Αν πραγματικά καθαρίσουμε την Ευρώπη, φανταστείτε τι θα γίνει πάρα πολλές και θέσεις εργασίας στην πορεία αυτή. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα, σχεδόν. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ευθυγραμμίσουμε την ταυτότητά μας με τον καθαρό αυτό κόσμο. Δεν θα ζητάμε κάτι, δεν θα πετούμε, αλλά θα δημιουργούμε κάτι νέο και ε, εύθραυτο και όμορφο. Αυτά είχα να πω. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ συγκεκριμένα θέματα έθεσες. Αλλά πίσω τους υπάρχουν και όνειρα. Είναι πολύ σημαντικό το όνειρο να συνδέεται από συγκεκριμένη εφαρμογή. Υπάρχουν ερωτήσεις και σχόλια στα μέλη του ακροατηρίου μας, αλλά ας πάμε στον τοίχο των tweet. Όπως βλέπετε, πολλά tweet και πολλές απευθείας ερωτήσεις στον ομιλητή. Οπότε σας καλούμε να απαντήσετε απευθείας στις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μερικές ερωτήσεις και για τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Ερώτηση από την εκδήλωση Σοφία. Πότε θα αισθανθούμε το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών πολιτών και πόσο θα κρατήσει η διαδικασία. Επίσης ένα tweet από την Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών γιατί μειώνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ευρωπαϊκά όργανα τη συμμετοχή των πολιτών μόνο μέσω τη Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλία των Πολιτών. Και πολλοί που στέλνουν ποιήτε ενδιαφέρονται για δικαιώματα μειονοτήτων. Ερώτηση από το γραφείο του Κοινοβουλίου στο, στην Πολωνία. Πώς θα συμμετάσχουν ε, οργανώσεις εθνικών μειονοτήτων στι εκδηλώσει αυτέ Και πολλέ ερωτήσει για το θέμα των Ρώμα. Πώ θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των Ρώμα και των ε, πληθυσμών του ταξιδιού και πολλή δραστηριότητα των tweet για το θέμα των νέων. Από όλα τα γραφεία του Κοινοβουλίου έχουν αποσταλεί ερωτήσεις. Για παράδειγμα στο γραφείο του ε, διαμεσολαβητή για το Πεδεμόντιο. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στις επόμενες ευρωεκλογές από το γραφείο του Κοινοβουλίου στην Ολλανδία. Πώς θα ενθαρρύνουμε και αυτούς ε, που δεν έχουν ακόμη δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των ενωσιακών πολιτικών. Από τη Σουηδία μας ρωτάνε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η ανεργία των νέων. Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό η Ένωση. Και τέλος, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, ένα tweet ε, από το γραφείο του Κοινοβουλίου στην Πορτογαλία για την νεολαία. Δεν θα έπρεπε να ανησυχεί η Ευρώπη για τη βελτίωση της εκπαίδευσης για να υπάρξει μια πιο ενωμένη ευρωπαϊκή ηθαγένεια, πιο ενιαία. Και πολλέ άλλε ερωτήσει για παρόμοια θέματα. Ωραία, εδώ το κοινό παρακαλώ. Είχατε ένα σχόλιο κυρία μου. Μαργαρίτα Άλβεν, είμαι ευρωβουλευτή πράσινη από τη Δανία. Είμαι συντονίστρια της Επιτροπής Αναφορών. Μία παρατήρηση για την πρωτοβουλία των πολιτών που απαντάει και σε κάποιες ερωτήσεις. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο Επίτροπος κ. Σεύκοβιτς στην προσπάθειά μας να υπάρξει αξιοπρεπής αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλειών πολιτών. Να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση. Οργανώνουμε ακροάσεις. Η Επιτροπή Αναφορών θα είναι η Επιτροπή που θα ε, προσπαθήσει να διασφαλίσει υψηλού επίπεδου συμμετοχή της Κομισιόν και τις ε, καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στους πολίτες ότι θα πάρουμε τις αποφάσεις που μας προτείνουν, αλλά να τεθεί ως θέμα στις συζητήσεις που κάνουμε. Είναι σημαντικό αυτό και ελπίζω η δική μας πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να ε, αντιμετωπιστεί καλύτερα από ορισμένες άλλες ε, που έχει οργανώσει η Κομισιόν. Και κάτι για τις ε, κλινικές δοκιμές. Συγχαίρω τον διαμεσολαβητή για την εργασία του για το θέμα αυτό, αλλά σας προειδοποιώ. Προέρχομαι από μια βόρεια παράδοση διαμεσολαβητών. Αυτό που μας απειλεί είναι ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχει τώρα μια τάση ε, δικοματικής ε, διακυβέρνησης ε, των πρωτοβουλειών μας. Και οι διαμεσολαβητές επίσης να προέρχονται από αυτά τα δύο κόμματα. Ανεξάρτητα από το πόσο εξαιρετικοί υποψήφοι μπορούν να υπάρχουν. είμαστε, εγώ προέρχομαι από την βόρεια παράδοση και εσείς κύριε Διαμαντούρε προέρχεστε από αυτήν την νότια παράδοση. Δεν έχει τίποτα να κάνει η σκέψη σας με τη χώρα προέλευσή σας. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η επιλογή των διαμεσολαβητών να μην είναι θέμα ε, μικροκομματικό. Θα πρέπει να υπάρχει αμεροληψία στον τρόπο επιλογής του διαμεσολαβητή, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το θεσμό. Είναι ο μόνος θεσμός που είναι έξω από το πολιτικό παιχνίδι μέχρι τώρα και κάνω έκκληση, παρακαλώ, να διατηρηθεί αυτή η παράδοση αντικειμενικότητα του διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Μπέρνς. Κάποιες ερωτήσεις βέβαια είναι αναμφίβολα και αναπόφευκτα πολιτικές. Αλλά παρακαλώ να ακούσουμε και μία άλλη ε, ομιλία. Ερώτηση μάλλον. Ρονόμπλασχερ από το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, το ΣΥΦ και πρώην Ευρωβουλευτής εδώ. Φαίνεται καθαρά ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αλλάζει μέθοδο. Και είναι εντύπωσή μου μετά από όσε περιπτώσει άκουσα σήμερα ότι αλλάζει και μέθοδο αλλά ίσω και το στόχο τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση ε, και φαίνεται ότι αποδίδεται ένα περισσότερο ανθρώπινο χαρακτήρα, περισσότερο ανθρώπινη Ευρώπη. Ε, και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τους πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών να μου απαντήσουν ε, τι διάσταση θεωρούν ότι η μέθοδος bottom-up αντί για top-down μπορεί να δώσει σε παρόμοιους στόχους όπως αυτούς που έχουν εκείνοι και εμείς σαν άνθρωποι επισημεριζόμαστε. Ο Άλμπερ Σβάιτσερ έδωσε ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα δεν είναι και το καλύτερο μέθοδος για να αλλάξει τα πράγματα αλλά είναι η μόνη. Και εδώ βλέπουμε στην Εσθονία αυτό. Αυτό το παράδειγμα το ακολούθησαν και στο Κωσυφοπαίδιο, που αλλού δεν θυμάμαι, Βοσνία νομίζω. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η τοπική δράση ενέργεια πώς μπορεί να βοηθήσει για τους στόχους αυτούς και πώς όλα αυτά μπορούν να συνοματωθούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ωραία. Μήπως ο Επίτροπος θέλει να απαντήσει πρώτος. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σεύκοβιτς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, του Twitter και των συμμετεχόντων εδώ στην αίθουσα. Πρώτη ερώτηση. Πότε θα αισθανθούμε τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών Πολιτών. Μα νομίζω ήδη τα αισθανόμαστε. Βλέπουμε από τη συζήτηση μας σήμερα, από τις συζητήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή από τη στιγμή που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών ότι υπάρχει μια νέα διάσταση συμμετοχικής δημοκρατία στην Ένωση. Μιλήσαμε για την απευθεία συμμετοχή, την απευθεία προσπάθεια επίδρασης ε, στην νομοθεσία. Και είναι πρώτη φορά που τα αναφέρουμε τα θέματα αυτά με τόσο συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή, γίνεται η Ευρώπη πολύ πιο ανθρώπινη. Και αυτό χρειαζόμαστε ιδιαίτερα τώρα στην τόσο δυσχερή συγκυρία. Τώρα, τι διαδικασίες και τι χρονοδιάγραμμα έχουμε μπροστά μας. Ξέρετε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το λογισμικό, γι' αυτό παρετάθη από την Κομισιόν η περίοδος κατά την οποία μπορούσαν να συλλεγούν υπογραφές. Έτσι λοιπόν, ε, το Νοέμβριο θα λήξει η μονοετής ε, περίοδος. Μετά θα χρειαστούν ε, δύο εβδομάδες περίπου τα κράτη-μέλη για να ελέξουν τις υπογραφές και μετά υπόσχομαι στην κυρία Όκεν ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να αντιμετωπίσουμε όλες τις πρωτοβουλίες με σωστό τρόπο. Υπόσχομαι λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει συνάντηση υψηλού επίπεδου μεταξύ των οργανωτών και των αρμοδίων επιτρόπων ή γενικών διευθυντών και ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι θα παίξει τον ρόλο του, θα οργανώσει όπως ακριβώς αρμόζει την ακρόαση. Γιατί είναι σημαντικό όχι μόνο να μπορούν οι διοργανωτές να μας εξηγήσουν την πείρα τους, να παρουσιάσουν το θέμα τους, αλλά να γίνουν συζητήσεις όπου θα δούμε διάφορες οπτικές γωνίες για τις προτάσεις, όπου θα υπάρξει επεξεργασία, όπου θα προκύψουν κατευθυντήρε γραμμέ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να κάνει τι ανακοινώσει για το πώ θα αντιμετωπιστούν οι πρωτοβουλίε. Αλλά ήδη σήμερα το διαπίστωσα. Και επίση το Σώμα των Επιτρόπων μου υποβάλλονται ερωτήσεις από τους συναδέλφους μου όσο προχωρούν οι πρωτοβουλίες, όσο διαπιστώνουμε πόσο στηρίζονται από τους πολίτες, ε, τι θέματα συγκεκριμένα περιέχουν. Ήδη επηρεάζουν τη συζήτηση που κάνουμε στην Επιτροπή επηρεάζουν την εργασία των επιτρόπων. Γίνεται λοιπόν ακουστή η φωνή των πολιτών. Θέλουμε να τους κινητοποιήσουμε. Στο μέλλον θα υπάρξει ακόμη περισσότερο η εξέλιξη αυτή. Διαπιστώσαμε τι ρόλο παίζουν και οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να κινητοποιήσουν τους πολίτες και τι μηνύματα μας στέλνουν. Το είδαμε, ε, το είδαμε και για μερικές διεθνείς συμφωνίες, το βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται η δημοκρατική συνειδητότητα, αλλάζει η νοοτροπία των πολιτών. Βλέπουμε πόσο, σε πόσο μεγάλο βαθμό κινητοποιούν τους πολίτες. Όσο πιο εύχριστο είναι το σύστημα, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα, όσο περισσότερο αξιοποιούμε το ψηφιακό θεματολόγιο, όλα αυτά, όλη αυτή η ηλεκτρονική δημοκρατία σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνουμε αποφάσεις αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το θεματολόγιο. Τα θέματα των Ρώμα και των νέων, μια λέξη μόνο. Ξέρετε, είμαι Σλοβάκος. Όπου υπάρχει σημαντική μειονότητα Ρώμα, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα θέματα Ρώμα αντιμετωπίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χρειαστήκαμε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα ε, που περικλείεται από εθνικά σύνορα. Πρέπει να ε, υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Πρέπει να μάθουμε ο ένας από τις βέλτιστες πρακτικές του άλλου. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που υπάρχει διαδικασία μιας ε, ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρώμα και επίσης απέτηση κάθε κράτος μέλος να έχει σαφή εθνική στρατηγική για να βελτιωθεί η ζωή των Ρώμα και οι στρατηγικές αυτές θα αποτιμηθούν συλλογικά είναι πολύ σημαντικό αυτό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Ρώμα να αντιμετωπίσουν τις δυσχέριές τους. Και τονίζω ότι η Επιτροπή το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά. Οι νέοι αντιμετωπίζουν ε, τρομερές δυσχέρειες, πρωτόγνωρες δυσχέρειες. Η γενιά αυτών των νέων είναι η καλύτερα εκπαιδευμένη και καταρτισμένη γενιά Ευρωπαίων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όμως υποφέρουν από το μέγιστο μεταξύ των άλλων κατηγοριών πληθυσμού ποσοστό ανεργίας. Τι να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Να βελτιώσουμε το πρόγραμμα σπουδών στα πανεπιστήμια, να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να βοηθήσουμε και τώρα αμέσως τους πολίτες μας για να μην υπάρξει χαμένη γενιά στην Ένωση. Τι προσπαθεί να κάνει η Ένωση πέρα από τις ήπιες εξουσίες που έχουμε ως Ένωση, ως Επιτροπή, γιατί ξέρετε ότι πολλά θέματα που αφορούν τον κοινωνικό τομέα για την εκπαίδευση είναι θέματα αρμοδιότητας εθνικών κρατών. Έχουμε δημιουργήσει ομάδες δράσης, θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους, ομάδες δράσης ιδίως στις χώρες που έχουν πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, για να αξιοποιηθούν αυτές οι πιστώσεις, ούτω ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Έχει λειτουργήσει, θα αποτιμήσουμε το πόσο είναι αποτελεσματικό και σας διαβεβαιώ ότι με βάση τις νέες πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές όπου έχουν δεσμευθεί έξι δις για αυτές τις πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Ελπίζω φυσικά όλα αυτά να γίνουν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να έχουμε μόνιμα αποτελέσματα και όχι μόνο παροδικά. Ο Πρόεδρος. Μας μένουν μόνο 20 λεπτά. Θα ήθελα να δοθούν ώστε να τον περισσότερες απαντήσεις, άρα παρακαλώ ώστε να τον συντομότερες απαντήσεις, παρακαλώ για να έχουμε πολλές. Να πάρει το λόγο η Αν Μάρη γιατί τέθηκε ένα ερώτημα το μπουινό για τις διαστάσεις που πρέπει να έχει αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Bottom up. Δύο απαντήσεις ε, το πώς επηρεάζεται η κατάσταση μετά από αυτή την πρωτοβουλία μας γιατί είμαστε στο κεντρικό σημείο. Δεν μπορούμε να δούμε ακόμα τις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα θα πρέπει να δοθούν ε, είτε στο χαρτί είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτές οι αναφορές και με επικύρωση ας το πούμε έτσι από τις εθνικές αρχές και να δοθούν αυτές στην Επιτροπή και νομίζω ότι έχει δύο, μάλλον τρεις μήνες διαθέσιμο χρόνο για να απαντήσει και μόνο από την χρονική αυτή στιγμή, τουλάχιστον για τη δική μας τον πρωτοβουλία, για το δικαίωμα στο νερό, θα δούμε εάν η Επιτροπή θα δεχτεί να προχωρήσει και να νομοθετήσει, είτε θα απορρίψει την πρωτοβουλία αυτή και όπως η Ιζαμπέλ Ντιρά μας το είπε πριν από λίγο τότε, ό,τι δεν μπορούσε να γίνει σε επίπεδο επιτροπής, τότε θα πρέπει να λεφθεί σαν προσπάθεια σε επίπεδο κοινοβουλίου. Και συνδυάζει έτσι την την ε, απόψη του Μπότονα από το κάτω προς τα πάνω και θα πρέπει να δούμε ότι αυτή πάντως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει και να ανέβει προς τα πάνω αυτή η ιδέα. Για τον τρόπο τώρα για την οικοδόμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πρωτοβουλίας αυτής για το δικαίωμα στο νερό. Έχουμε ορισμένες δεσμεύσεις σε τοπικό επίπεδο με τους εκλεγμένους, δημοτικούς συμβούλους κλπ, διάφορες ομάδες και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί μια διάσταση ανθρώπινη, σαν θεμελιώδες δικαίωμα. Έχουμε τη χάρτα αυτή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία και έχει ενταχθεί στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας και πάνω σε αυτό, σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να δηλώσουμε και εμείς ότι συμμετέχουμε και εδώ ολοκληρώνω θα μπορούσε και μέσω αυτών των πρωτοβουλειών των πολιτών να δοθεί η δυνατότητα για μια επανεξισορρόπηση ανάμεσα στα όσα γίνονται και μας τα γενικά έτσι ε, σχεδόν ε, στα κρυφά από εκείνους που ασχολούνται και εδώ μιλάω για τη δραστηριότητα των ομάδων πίεσης, τα λόμπις ξέρουμε ποιο είναι το βάρος που έχουν στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς από τη στιγμή εκείνη που οι ενέργειε των πολιτών, των ενεργών, όπως το, θα το ήθελε και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και μέσω ίσως και ορισμένων αφελών αλλά και ιδεαλιστών θα μπορέσει να δοθεί η διάθεση στον άγνωστο πολίτη να καταβάλει μια προσπάθεια να συμμετάσχει και να πει από τη στιγμή που με ακούν ε, και όχι μόνο με ακούν αλλά και κάνουν αυτά που τους λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε γρήγορα στο Χάινορ, γιατί υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις, κυρίως για, ε, από νέους. Και στα βίντεο που μας δείξατε ήταν πολύ νέοι, κάτω από την ηλικία της, που ψηφίζουν. Όπως ακούσαμε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κάτω αλλά και από αλλού, η ερώτηση είναι πώς κάνεις τους νέους να συμμετέχουν. Εσύ το έκανε με επιτυχία. Και πώς του κινητοποιείς, κυρίως του χρόνου, αυτούς που μπορούν να ψηφίσουν, πώς τους κάνεις να αναγνωρίσουν ότι φέτος είναι το έτος των πολιτών και του χρόνου είναι η χρονιά που θα ψηφίσουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς να τους κινητοποιήσω να ψηφίσουν, δεν έχω ιδέα. Αν θες να αγγίξεις τους ανθρώπους αυτούς, Πρέπει να είσαι ειλικρινής. Αυτό το λες εύκολα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι, έχουν συνηθίσει να λένε αυτά τα οποία σκέπτονται. Δεν έχουν, ε, δεν έχουν γνωρίσει τις εποχές που εμείς γνωρίσαμε. Είναι δηλαδή θέμα γλώσσες, λέει ο Προεδρεύων. Είναι θέμα ε, του να ακούς τι λέει η καρδιά σου και να λες τι πιστεύεις. Δεν είναι θέμα πολιτική, πολιτικής. Ποιες λέξεις χρησιμοποιείς. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις δεν είναι θέμα λέξεων, είναι θέμα του τι αισθάνεσαι. Και πάντοτε με εντυπωσιάζει ότι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι μπορούν να παίξουν με τα λόγια για να κάνουν εντύπωση. Σήμερα αυτό δεν είναι δυνατόν. Ερώτηση. Πώς μπορείς να κάνεις τους νέους και τους νέους ψηφοφόρους να πάνε στην, ε, να ψηφίσουν. Ε, ομά, την έχουμε πατήσει. Και ας καθαρίσουμε τα πράγματα όλοι μαζί. Αυτή είναι η ουσία. do we have any more... Ερώτηση. Έχουμε περισσότερα. άλλα tweet. Δύο άμεσα ερωτήματα, γιατί πρέπει να μην καθυστερήσουμε και πολύ. Από το γραφείο του Κοινοβουλίου στην Πολωνία, μια ερώτηση προς τον Ράινερ. Από όσο έχει από όσο γνωρίζεις, πόσο μπορούμε να συμμετέχουν ε, αποτελεσματικά πολιτικοί στις τοπικές πρωτοβουλίες. Και ερώτηση προς τον ε, διαμεσολαβητή. Το Γραφείο της Ρουμανίας θέλει να μάθει πώς ε, συνεργάζεστε με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Άλλη ερώτηση από την αίθουσα. Είμαι ο Άντρες Γκόμπινς από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρευρεθώ και να συμμετάσχω στη συζήτηση ταυτόχρονα με τις εθνικές συζητήσεις. Το εθνικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να γίνονται συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Αυτό βεβαίως αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για όλους. Ερώτηση. Μιλά... Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, που αποτελεί ευκαιρία για να επιτευχθούν συγκεκριμένα πράγματα. Ίσως εσείς και ο Επίτροπος θα μπορούσατε να μας αναφέρετε παραδείγματα ε, πρωτοβουλειών που αναλάβατε για να επικοινωνήσετε εσείς από πλευρά σας καλύτερα με τους πολίτες. Μπορείτε να μας αναφέρετε συγκεκριμένες περιπτώσεις πραγμάτων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. Ευχαριστώ. Μια άλλη ερώτηση. Είμαι η Ρέτσολ Χάμζη που εργάζομαι για το παρατηρητήριο της ε, Εταιρικής Ευρώπης και θέλω να επισημάνω το εξής. Η μία πλευρά κάνει τους, αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν για την πολιτική να ακούσουν για τους πολίτες και από την άλλη πλευρά μιλάμε για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτά τα οποία λένε. Όμως υπάρχει ενδιαφέρον από ε, συγκεκριμένα εμπορικά συμφέροντα, μεγάλες βιομηχανίες που παρακολουθούν μέσω ομάδων πίεσης. Είδαμε και το παράδειγμα του Thomas Λόγκριν στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Είδαμε παραδείγματα που για λόγους καριέρας και εμπορικούς λόγους η θετική πολιτική που είναι στο συμφέρον των πολιτών υπονομεύεται. Ερώτηση προς τον Επίτροπο. Τι, κάνει, τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει πολύ καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις φωνές των πολιτών σε σχέση με τις φωνές του εμπορικού κόσμου και προς τον διαμεσολαβητή. Αυτή τη στιγμή ε, έχετε δεχθεί ε, μια καταγγελία από τη δική μου και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το πώς θα ε, αντιμετωπίσει το θέμα των των συμφερόντων η Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαπλοκής, τι σκοπεύετε να κάνετε σε διαρθρωτικό ή πολιτιστικό τρόπο για να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην πολιτική. Φόρε, νομίζω ότι απευθύνθηκαν σε σένα αρκετές ερωτήσεις, μπορώ να σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Πάρα πολλές ερωτήσεις ε, μου απευθύνθηκαν. Θα κάνω κάτι που δεν είναι πολύ συμβατικό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συγκεντρώνοντας κάποια πράγματα μαζί και κατόπιν θα προσπαθήσω να αναφερθώ και σε κάποια από τα συγκεκριμένα ζητήματα αν έχουμε χρόνο. Θα επιλέξω ε, λεξούλες, ήχους. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε ε, για πράγματα τα οποία λέει γίνονται τώρα που μιλάμε ή υπάρχει και το εκ των κάτω προς τα άνω ή η ανθρώπινη διάσταση ή το να είμαστε ειλικρινείς. Αυτά ακούστηκαν. Αυτό το οποίο εκπροσωπεί κυρίως αυτή η εκδήλωση και η περσινή εκδήλωση είναι το εξής βλέπουμε μια ευνίδια σημαντική επίπτωση στην κοινωνία μας που προήρθε από την πληροφορική και τα κοινωνικά μέσα. Μια ταχεία αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου και το πώς ερχόμαστε σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Ακριβώς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή με την επαφή με 30 πόλεις οι οποίες υποβάλλουν ερωτήσεις. Και ευθύς είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης μαθησιακής καμπύλης που θα μας μετακινήσει σε μια άλλη κατεύθυνση στον τρόπο που ερχόμαστε σε επαφή μεταξύ μας και με τους πολίτες. Αυτό θέλω να το καταγράψω, να πω ότι ο διαμεσολαβητής πιστεύει ότι σε κάποιο βαθμό, εν, εν μέρη τουλάχιστον, έχουμε πιάσει το σφιγμό αυτού που γίνεται. Δεν θέλω να, καφ, να ούτε να συγχαίρω τον εαυτό μου, αλλά να πω ότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα η οποία εμφανίζεται ταχύτητα και θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε ότι εσείς και εμείς, γιατί ο διαμεσολαβητής είναι ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς και εμείς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα πράγματα. Και αυτό προσπαθεί να κάνει το γραφείο μου τα τελευταία 8 χρόνια και ελπίζω και η διαδοχή μου να το κάνουν αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Πράγματι, ο διαμεσολαβητής πολύ συχνά περιγράφεται ως το ανθρώπινο πρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Βεβαίως. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εσείς βεβαίως θα πρέπει να μας κρίνετε, να μας ε, και γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και αυτό πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε. Και βεβαίως όταν συμβεί αυτό θα έχουμε περισσότερες περιπτώσεις που θα κινούνται τα πράγματα εκ των κάτω προς τα άνω. Και ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαϊκές ε, Πρωτοβουλίες Πολιτών. Τώρα, να απαντήσω και σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα να ευχαριστήσω την κυρία Κουέν για τα σχόλιά της. Ως ο τρέχον διαμεσολαβητής δεν είμαι ε, σε θέση να μιλήσω για τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου μου, αλλά ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει εν τη σοφία το αυτό που έχει κάνει στο παρελθόν, ότι θα δώσει έναν καλό διαμεσολαβητή στο μέλλον και θέλω σε σχέση με αυτό να αναφέρω την παρουσία, μας, παρουσία εδώ ανάμεσά μας, τεσσάρων τουλάχιστον διαμεσολαβητών, είναι ο κύριος Σαμπό, εθνικός ε, διαμεσολαβητής της ε, Ουγγαρίας, κυρία Οράιλι της Ιρλανδίας, προηγουμένως ο κύριος Άλεξ Μπρένινγκ της Ολλανδίας και επίσης έχουμε έναν υποψήφιο για τη θέση του διαμεσολαβητή, Μάρκες Γέγκερ, ένα ανώτατο στέλεχος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία για να εξασφαλίσουν ότι αυτός ο θεσμός θα συνεχίσει να προσφέρει στους πολίτες ό,τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα και στο μέλλον. Ποια είναι η σχέση του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή με τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρότερο δίκτυο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 18 χρόνια. Είναι ένα ένα δίκτυο που συγκεντρώνει όλους τους περιφερειακούς και εθνικούς διαμεσολαβητές ε, ε, κάθε ε, δύο χρόνια, μία χρονιά για τους εθνικούς και μία για τους περιφερειακούς. αυτό συντονίζεται από το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχουμε ένα ειδικό σημείο στην ε, ιστοσελίδα μας και έχουμε και μια καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα που απευθύνεται στους εθνικούς διαμεσολαβητές. Μπορείτε πάντοτε να πάτε στον εθνικό διαμεσολαβητή για να έρθετε σε εμά ή και από εμά για να στείλετε μηνύματα. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που επιτρέπει στους πολίτες να έρθουν σε επαφή με τους δύο διαμεσολαβητές σε εθνικό ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο διαμεσολαβητής ανησυχεί πολύ για τα δικαιώματα των μειονατήτων, για, κυρίως για τους Ρωμά, γιατί είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι, ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και ανησυχεί για τα, τα, με τα προβλήματα της νεολαίας. Επίσης, πρέπει να προσθέσω, ενδιαφέρεται και εμπλέκεται ενεργά στην υπεράσπιση δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει την πρώτη της σύμβαση με τα Ηνωμένα Έθνη και είμαστε τώρα στην πορεία δημιουργίας ενός μηχανισμού, ενός πλαισίου όπως το ονομάζουμε στην γλώσσα της γραφειοκρατίας, μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή στην πράξη αυτής της συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών επί εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γραφείο του Διαμεσολαβητή είναι ένας από τους τρεις συμμετέχοντες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το θέμα πάρα πολύ ενεργά. Επίσης υπάρχουν πολλές καταγγελίες και δρούμε σε πολλούς τομείς που αφορούν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, γιατί ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτικός για τα ε, κράτη-μέλη που εφαρμόσουν το ενωσιακό δίκαιο και δεσμευτικό για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπάρχουν απόλυτες ε, νομικές εγγυήσεις για τα δικαιώματα πάσης φύσεως μειονοτήτων. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας όπου είναι σε επιφυλακή ο διαμεσολαβητής και όπου συμμετέχει πολύ ενεργά. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα από το παρατηρητήριο των ε, εταιρικών ε, ε, υποθέσεων. Πρέπει να πω ότι η υπόθεση αυτή βρίσκεται εν εξελίξη, δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε. Από την ώρα που θα ολοκληρωθεί, θα καταγραφεί και βεβαίως ο διαμεσολαβητής είναι σε επιφυλακή για την ε, προστασία των νομίμων των αρχών του, της, ενόμου τάξεως, του κράτους δικαίου, στην πράξη το, σε θέματα πρακτικής, δια, διαπλοκών και, και αλλά πρέπει πρώτα να μελετήσω τι συμβαίνει πριν να αποφασίσω και αυτό δεν το έχω ακόμα κάνει. Γι' αυτό λέγεται παρουσία του υπευθύνου επιτρόπου. Ακριβώς εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όταν θα έχω προχωρήσει περισσότερο θα μπορέσω να πω κάτι παραπάνω. Ιδάλλως θα είμαι άδικος και στις δύο πλευρές και αυτό δεν θα ήθελα να το κάνω. Ε, παραδείγματα συγκεκριμένων πρακτικών. Θεωρώ ότι ο κύριος Γκέτσεκ σας έδωσε ένα πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που καταφέραμε να αντιστρέψουμε μια μακρά πολιτική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που πλέον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα των κλινικών δοκιμών. Να σας το πω ως εξή. Πριν από 10 χρόνια, όταν ήρθα στην Ένωση, υπήρχαν 10 αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή στιγμή είναι 43. Πολλοί από αυτούς είναι ρυθμιστικοί δραστηριότητες οργανισμοί, των οποίων οι δραστηριότητες αγγίζουν πραγματικά την καθημερινή ζωή των πολιτών των κρατών μελών. Τρόφιμα. Φάρμακα περιβάλλον, σύνορα, χημικές ουσίες. Όλα αυτά αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών και όλα αυτά είναι στο πεδίο τη αρμοδιότητάς μου. Έχω επισκεφθεί όλους αυτούς και έχω ξεκινήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αυτοί τηρούν τις ε, υποχρεώσεις του, δυνάμει του, του ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, του ενωσιακού δικαίου και ότι έχουν συνέστηση της ανάγκης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου ώστε να μπορούν οι ε, πολίτες να γνωρίζουν και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά του. Έτσι λοιπόν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ένας από τους οργανισμούς. Η πρωτοβουλία μου αφορά όλους τους οργανισμούς και υπάρχουν 18 ή 19 που έχουν καλυφθεί. Όλοι σημαντικοί εκτός του Οργανισμού Τροφίμων δεν μπόρεσα να επισκεφθώ την Πάρμα Αυτά είναι όλα επιπλέον παραδείγματα. Τελικό παράδειγμα, τα τελευταία 10 χρόνια ο διαμεσολαβητής έχει σταθερά προσπαθήσει να προωθήσει τα όρια της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, του να είναι κανείς υπόλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι δημοσιεύσαμε μια έκθεση και αναφέραμε 82% ε, συμμόρφωση από πλευρά όλων των οργανισμών στη συστάση μας. Δεν ξέρω, οι πολίτες θα κρίνουν αν αυτό είναι αποδεκτό επίπεδο ή όχι. Θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος πελάτης μας εντός εισαγωγικών, και δεν μου αρέσει ο όρος αυτός, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο, τρίτα των καταγγελιών που ε, έρχονται είναι αφορούν την Επιτροπή. Παρουσία του αρμοδίου Επιτρόπου θα πρέπει να πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καλή, αλλά είναι τα προβληματική διοίκηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. υπαλλήλου. 36.000 από είναι πολύ καλή, αλλά είναι τα δύο τρίτα τη συνολικη διοικηση ευρωπαικη ενωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου 55.000 υπαλληλου 36.000 από αυτου είναι υπάλληλοι τη ευρωπαικη Επιτροπής. Άρα είναι αναπόφευκτο για αυτούς προ εκεί να απευθύνονται τα περισσοτερε καταγγελιε ομω πέρυσι ήταν 82%. Έχει αυξηθεί σταθερά αυτό ο αριθμό, αυτό το ποσοστό. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε σιγά και σταθερά να προωθήσουμε τα όρια της καλής διοίκησης. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το πώς προωθεί κανείς μια νοοτροπία για την εξυπηρέτηση. Η Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση να πιστεύει ότι το κράτος βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετεί τους πελίτες και όχι αντιστρόφως. Αυτά είναι αυτά τα οποία κάνει τα δέκα τελευταία χρόνια ο διαμεσολαβητής. Αν μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα, έχετε μισό λεπτό λέει ο Προεδρεύων. Μία ερώτηση αφορούσε το προφίλ που θα ήθελα να έχει ο μελλοντικό διαμεσολαβητής. Απαντώντας λέω ότι όλα όσα σας είπα ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία δέκα χρόνια σας δίνει την σύνθετη εικόνα του των δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος μεσολαβητής, ο οποίος πιστεύω θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, χτίζοντας στις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό και να προωθηθεί ακόμα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ε, κύριε Διαμαντούρα, που ε, φτάσετε στο τέλος της δεκαετούς θητείας σας ως διαμεσολαβητής οποιοδήποτε θα σας διαδεχτεί έχει δυσχερές καθήκον και δεν θα το ευχόμουν σε, σε κανέναν. Κανείς δεν θα λένε στα παπούτσια σας τα οποία λέει ο κ. Διαμαντούρος είναι μέγεθος 43. Υπάρχουν λοιπόν τα γραφεία του Κοινοβουλίου, υπάρχουν οι, ε, όσοι μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Αυτό το τρίωρο για μένα ήταν ιδιαίτερα υποφελές ως ε, συντονιστής ε, ε, προγραμμάτων του Euronews. Συνήθω έχω μόνο 10 λεπτά, όπως θα έχω και σήμερα το απόγευμα, για το θέμα της φοροδιαφυγής. Σήμερα όμως είχαμε 3 ώρες. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν πολλές πλευρές των θεμάτων αυτών. Θα τις συζητήσουμε και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διοχετεύσουμε και τον θυμό, αλλά και τη δημιουργικότητα και τα όνειρα των πολιτών είτε μέσω του διαμεσολαβητή, είτε μέσω αναφορών, είτε μέσω των πρωτοβουλειών βάσης που εσείς διοργανώνετε. Φέτος είναι το έτος των πολιτών και ε, του χρόνου που θα έχουμε ευρωεκλογέ. Πρέπει να προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα γιατί πρέπει να υπάρξει υψηλή συμμετοχή. Αν δεν υπάρξει θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη αποτυχία για την Ένωση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγάλη ενεργητικότητα και Νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον που όλοι πρέπει να προωθήσουμε και αυτό προωθώ και εγώ σε Ευρωπαίους πολίτες. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να του χρόνου.